Okay, thank you, gentlemen of the press. Ευχαριστώ κύριοι δημοσιογράφοι. Πρέπει όμως να αρχίσουμε. Καλημέρα κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Καλωσορίζω τον υποψήφιο επίτροπο Κάρολο Ντεχούχτ. Τονίζω ότι ποια είναι η σημασία αυτής της συνεδρίασης. Είναι ζωτική στιγμή του ορισμού των επιτρόπων με έλεγχο από τους πολίτες. Και έτσι εκφράζονται οι αρχές του δημοκρατικού ελέγχου που μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει στο διακυβερνητικό σύστημα της Ένωσης. Η σημασία τέτοιων ακροάσεων έχει αυξηθεί επειδή η συνθήκη της Λισαβόνας έχει δώσει στην Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο αυξημένες δικαιοδοσίες και ευθύνες για τη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να γνωρίζει τι μπορεί να αναμένει από τον μελλοντικό εμπορικό επίτροπο. Μέλλοντα, μέλλοντα. Γιατί έχουμε νομοθετικές συνυπευθυνότητες και είμαστε το μόνο εκλελεγμένο όργανο από τους πολίτες. Φυσικά αυτό, ο έλεγχος δηλαδή, είναι κάτι πολύ θετικό και εξ ονόματος των μελών της Επιτροπής μας δηλώνω ότι προσβλέπουμε με μεγάλες προσδοκίες στην άσκηση αυτών των καθηκόντων. Αρχίζω υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με αυτά που έχουμε αποφασίσει και με αυτά που λέει ο κανονισμός το Κοινοβούλιο εξετάζει τις γενικές ικανότητες του υποψηφίου, την προσωπική του ανεξαρτησία, καθώς και τις γνώσεις του θέματος του και τις επικοινωνιακές του ικανότητες ο υποψήφιος έχει ήδη υποβάλει γραπτός απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις και οι απαντήσεις του έχουν διανεμηθεί σε όλες τις γλώσσες στα μέλη. Σύμφωνα με τον κανονισμό επίσης λάβαμε από την Κομισιόν τα στοιχεία που δήλωσε ως συμφέροντα ο υποψήφιος. Και τώρα τα διαδικαστικά. Υπάρχει διερμηνία σε 22 γλώσσες από και προς και θα ήθελα να σας παρακαλέσω για να βοηθήσετε τους ερμηνευτάς και τα ερμηνευτρίας να μην μιλάτε πολύ γρήγορα για να προλαβαίνουν να μεταφράζουν. Επίσης αναμεταδίδεται από τον ιστότοπο του Κοινοβουλίου η, δια... η συνεδρίαση και θα παραμείνει και στα οπτικοακουστικά πρακτικά. Σημειώστε παρακαλώ ότι εκτός από την αίθουσα αυτή υπάρχει και πρόσθετη αίθουσα στην οποία να μεταδίδεται η συνεδρίαση στο α5γ3. Η ακρόαση θα έχει την εξής δομή. Έχουμε τρεις ώρες ακριβώς. Τα έχετε στους φακέλους σας. Ο υποψήφιος στην αρχή θα κάνει αρχικές δηλώσεις το πολύ 10 λεπτών και μετά ερωτήσεις για 2 ώρες και 45 λεπτά σύμφωνα με την αρχή του επιτραπεζίου τένις, της επιτραπεζίου αντισφαιρίσεως ή πινκ-πονγκ. Στην αρχή οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων με πεντάλεπτες παρεμβάσεις, άρα μονόλεπτη ερώτηση, απάντηση του κυρίου Ντεχούχτ, δίλεπτη, επόμενη συμπληρωματική ερώτηση ενός λεπτού και συμπληρωματική απάντηση δύο λεπτών, σύνολο πέντε για τον καθένα. Για τα τετράλεπτα που έχουν χορηγηθεί, ερώτηση 1, απάντηση 1, αντερώτηση 1, ανταπάντηση 1. Ο χρόνος ομιλίας των μελών περιορίζεται αυστηρά στο 1 λεπτό. Οι ερωτήσεις και οι συμπληρωματικές πρέπει να τίθενται από τον ίδιο άνθρωπο και να αφορούν αυτά που απαντάει ο υποψήφιος. Οι συμπληρωματικές ερωτήσεις δηλαδή δεν μπορούν να θίξουν διαφορετικά θέματα από το προηγούμενο. Και ο πρόεδρος θα απαγορεύει την υποβολή συμπληρωματικών και διαφορετικών ερωτήσεων. Θα είμαι αυστηρότατος στο σεβασμό του χρόνου ομιλίας. η γραμματεία προσπάθησε να έρθει σε επαφή και με τους μη εγγεγραμμένους αλλά δεν το κατάφερε και γι' αυτό τα πέντε λεπτά για εκείνους έχουν προσθεθεί στον γενικό συνολικό χρόνο για τις τελικής απαντήσεως του υποψηφίου και του Προέδρου μας, εμού δηλαδή του ιδίου. Ο τελικός χρόνος λοιπόν για τις δύο αυτές τελευταίες δηλώσεις γίνεται 10 λεπτά αντί για 5 που ήταν αρχικά. Θα γίνει και μία συνέντευξη τύπου αμέσως μετά. Αυτά είναι τα διαδικαστικά και αρχίζει τώρα η ακρόαση. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντεχούχτ για τις αρχικές του δηλώσεις και την παρουσίαση. Δέκα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι για την ευκαιρία που έχω σήμερα να σας συστηθώ στην Επιτροπή σας παρουσία εκπροσώπων και άλλων ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών διεθνούς ε, αντικειμένου και να σας ε, εκθέσω τις απόψεις μου για το διεθνές εμπόριο. Ελπίζω δε να είναι η πρώτη και όχι η τελευταία σειρά συζητήσεων που θα ακολουθήσουμε. 15 χρόνια εμπειρία έχω ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βουλευτής και στη συνέχεια διατέλεσα επίτροπος για θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας και έχω πραγματικά μεγάλη εμπειρία και μπορώ να διασφαλίσω το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύεται ε, σε θέματα εμπορικής νομοθεσίας και εμπορικών συμφωνιών και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ γνωρίζω τον κόσμο του Διεθνούς Εμπορίου ως υπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου. Έχω συλλέξει εμπειρία ακριβώ σε τέτοια θέματα εμπορίου και αναπτυξιακή συνεργασία και διεθνών σχέσεων γενικότερα. Έχω εκπροσωπήσει το Βέλγιο σε υπουργικέ διασκέψεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε υπουργικά συμβούλια, αλλά και ε, στο Χονγκ Κόνγκ του ΠΟΕ το 2006 ε, και στη Γενέβη το 2008 στις υπουργικές αυτές ε, συναντήσεις. Επιπλέον ε, είχα ηγηθεί και μια σειρά αντιπροσωπιών ε, εμπορικού αντικειμένου σε 12 χώρες. Έχω λοιπόν συλλέξει την απαραίτητη εμπειρία και τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ένας διαπραγματευτής. Και ε, ως προβουλευτής και ως πολιτικός στο Βέλγιο έχω εμπειρία στο πώς φυριλατούνται οι συνασπισμοί κομμάτων και πώς γίνονται διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι σημαντικό και στην καθημερινή πολιτική και την ευρωπαϊκή και τη βελγική. Έρχομαι τώρα στα αγγλικά γιατί αυτά τα είπα στα ολλανδικά. Το χαρτοφυλάκι όμως ανέκαθεν ήταν ε, ευκαιρία για ανάπτυξη και στην Ευρώπη και αλλού. Ακόμα και σήμερα είναι μια ευκαιρία για να βγούμε από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση. Εγώ είμαι ένθερμος υποστηρικτής ε, παγίως ε, της εμπορικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του ελευθερού εμπορίου χωρίς να πιστεύω ότι είναι αυτός σκοπός με τρόπο απλουστευτικό. Θα πρέπει το ελεύθερο εμπόριο να είναι στην υπηρεσία της ευημερία, της ανάπτυξης και να έχουμε τελικά όφελος για όλα τα μέρη. Είναι σημαντικός μοχλός μεταξύ άλλων μέτρων για προωθούνται ευρωπαϊκές αξίες όπως είναι η φοροσανάπτυξη, ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιπλέον ε, η διάνοιξη των ιδίων μας των αγορών δημιουργεί καινοτομία ε, και πρόοδο στη χώρα μας και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στο ε, διεθνέ εμπόριο σε αντίστοιχο ανοιχτό δρόμο. Θα πρέπει να ηγούμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το παράδειγμά μα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δεχόμαστε αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ ή προστατευτικέ από ε, άλλα κράτη. Γι' αυτό, απαντώντα στι γραπτέ σα ερωτήσει, επέμεινα ότι το εμπόριο θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία των ευρυτέρων στόχων πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε που είμαι μέλο Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο Ιούλιο έχω καταλάβει καλύτερα τα συστήματα ε, για το διεθνές συμπόριο και θα είμαι προσιλωμένο προ την κατεύθυνση αυτή με τη δική σα συνεργασία. Η ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου θα πρέπει να υποστηρίζει στεναρά τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε του κόσμου για να μπορέσουν να ενταχθούν ε, στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και να ε, αυξηθεί και το βιωτικό τους επίπεδο και να επέλθει κοινωνική πρόοδο στις χώρες αυτές. Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη, να σα αναφέρω τι εξή προτεραιότητε για την επόμενη πενταετία στο εμπόριο. Πρώτον, θα πρέπει να ενισχύσουμε και να διατηρήσουμε το πολυμερές σύστημα εμπορίου. Αυτό τον καιρό υφίσταται πιέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, Εμπορίου. Από το 2001 δεν έχει προχωρήσει ο γύρος διαπραγματεύσεων τη Τόχα. Ε, μιλούμε για συστήματα ε, πολυμερή, πολύπλευρα με διαφάνεια με ένα μηχανισμό διακανονισμό των διαφορών και είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτού του 20ου αιώνα. Ένα φόρουμ, ο ΠΟΕ, ε, ας πούμε, για να ε, ξεφύγουμε από την κλιμάκωση του προστατευτισμού για να λυθεί το περίφημο θέμα της διένυξης της μπανάνας που κρατούσε τόσο γερό στο παρελθόν. Είναι ένας τρόπος να ξεφύγουμε και στη σημερινή κρίση από το προστατευτισμό. Α μην ξεχνάμε ότι σε σύγκριση με του διεθνεί οργανισμού, όπου είναι το μεγαλύτερο και το πιο προχωρημένο ε, παράδειγμα παγκόσμια διακυβέρνηση που υπάρχει θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να επενδύουμε στην κατεύθυνση αυτή. Στη συνέχεια, να εμβαθύνουμε το εμπόριο και τις επενδύσεις και αυτό είναι συμπληρωματικό και όχι υποκατάστατο. Η Ινδία, ο Καναδά, η Λατινική Αμερική, η Ουκρανία, η Ευρωμεσογειακή είναι θέματα που θα κυριαρχήσουν μάλλον το επόμενη διετία ε, στις εργασίες μας, όπως και οι υπερχόμενες ε, συζητήσεις με τη Σιγκαπούρη και αναβάθμιση των εμπορικών μας σχέσεων με την Κίνα. Ε, όλα αυτά ανοίγουν σημαντικές αγορές που μετατοπίζονται ιδιαίτερα στην Ασία, αλλά σημαίνουν και βαθύτερη ένταξη και συνεργασία με τους γειτονές μας. Γνωρίζετε ότι επίκειται η συμφωνία με την Κορέα ε, και θα σας υποβληθεί προς έγκριση. Νομίζω ότι είναι καλή η συμφωνία αυτή και θα είναι προς όφελος της οικονομίας μας και προσβλέπω στη συζήτηση στην Επιτροπή σας και στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό. Επόμενο στόχο, οικονομική συνεργασία με άλλε ηγετικέ οικονομίε παγκοσμίω σε υψηλό επίπεδο και να μην αφήσουμε τα θέματα αυτά στα χέρια των ΗΠΑ και τη Κίνα. Το πρόβλημα με τις ΗΠΑ δεν είναι φραγμή στα σύνορα, αλλά πίσω από τα σύνορα, με διάφορους κανονισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου ε, ζήτησε ε, μια μελέτη για τις ε, συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε και τα ωφέλη που έχουμε από την άρση των τελωνιακών φαρμακών. Θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικού ντάμπινγκ κυριαρχούν ζητήσεις και η μη τελωνιακή φραγμή θα είναι προτεραιότητά μου στο Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο ε, που θα συμπροεδρεύω από ευρωπαϊκής πλευράς. Θα πρέπει επίσης να εντείνουμε το διάλογό μας με την Κίνα για τις ε, επενδύσεις και το εμπόριο καθώς το Πεκίνο καθίσατε όλο και περισσότερο πρωταγωνιστή στα παγκόσμια οικονομικά πράγματα. Ελπίζω να βελτιώσει τη διαφάνεια και να ανοίξει την αγορά της το εμπόριο και τις επενδύσεις ε, Κίνα και να συζητήσει και θέματα καθόδη όπως νομισματικά και ισοτιμίες. Στη συνέχεια θα πρέπει να οδηγηθεί σε επιτυχία η συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ. Ε, αυτές οι συμφωνίες δέχονται πολλές κριτικές και από τις χώρες εταίρους και από την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική των τελευταίων μηνών πάντα με στόχο ε, συμφωνίες που να συνάδουν και με του στόχου του ΠΟΕ και με την ανάπτυξη. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια νέα γενιά συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων στι 31 Δεκεμβρίου 2011 που λύγει το παρόν σύστημα. Και τέλο. Ακριβώ επειδή είναι δύσκολη οικονομικά η καιρή, θα πρέπει να βεβαιωθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι ευρωπαϊκέ εταιρείε ε, εισαγωγή, εξαγωγή ή ανταγωνιστέ άλλων θα πρέπει να έχουν δίκαιης μεταχείρισης και ε, να τη χάνουν συγγνώμη και να έχουν τις ευκαιρίες με άλλες. Στην πρόσβαση σε τρίτες αγορές. Επίσης, θέλω να ε, επιβληθούν και να χρησιμοποιούνται σωστά τα αισθήματα που έχουμε ε, για να προστατεύουμε το εμπόριο. να οδηγηθεί σε αίσιο πέρας ο γύρος της Δόχα και να δούμε πώς μπορούμε ε, με τις νέες αξίες που έχουμε για τις άμεσες εξένες επενδύσεις να ε, βοηθήσουμε και να βεβαιωθούμε ότι οι φυστάμενες συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών θα παραμείνουν σε ισχύ. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσουμε για μια νέα επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, σε επίπεδο νομοθεσίας και σε επίπεδο κρατομελών. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, αυτή βλέπετε ότι είναι μια πλήρης ε, ατζέντα, ένα πλήρης πρόγραμμα. Χρειάζομαι βοήθεια όμως για να το υλοποιήσω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να ε, ασκήσει πλήρω τι νέε αρμοδιότητε, συμπεριλαμβανομένε μια νέα συμφωνία πλαισίου μεταξύ των θεσμικών μα οργάνων. Και μπορείτε είστε βέβαιοι ότι θα συνεργαστώ και στην Επιτροπή σα και στην Ολομέλεια σε πλήρη διαφάνεια για το εμπόριο και θα σα δίνω πάντα τι πληροφορίε που χρειάζεται για να κάνετε τη δουλειά σα. Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντοτε, αλλά ε, θα δείτε ότι είμαι πάντα πρόθυμος να σας ακούσω και η πόρτα μου θα είναι πάντα ανοιχτή αν θέλετε να πούμε και σε λεπτομέρειες τις ερωτήσεις και απαντήσεις, αλλά η αφετηρία μου είναι να γνωρίσω ότι η Λισαβόνα χρειάζεται ποιοτική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Στα γαλλικά τώρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, στον χρόνο που μου δόθηκε δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω για όλα τα θέματα στα οποία άξιζε να αναφερθώ, α πούμε, η σχέση εμπορίου με την κλιματική αλλαγή ή το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω να τα θέσετε στις ερωτήσεις σας έτσι ώστε να μπορέσω να σας δώσω το πολιτικό μου όραμα για τα θέματα αυτά. Ε, επιτρέψτε μου τώρα να κλείσω με το εξή μήνυμα. Η εμπορική πολιτική είναι σίγουρα σημαντικός μοχλός της οικονομικής μας πολιτικής. Πλην όμως παραμένει στην υπηρεσία ευρυτέρων στόχων της κοινωνίας μας όπως είναι ο σεβασμός των κοινωνικών δικαιωμάτων, η καλή διακυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντο Πρόκειται λοιπόν για ένα κατεξοχήν πολιτικό ε, εργαλείο και θα πρέπει να ακούγεται και η πολιτική φωνή του Κοινοβουλίου με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντεχούχτα. Περνάμε στην πρώτη ομάδα των ερωτήσεων. Ξεκινάμε με τους συντονιστές τους ε, ε, της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου. Ξεκινάμε τον ε, κύριο Κάσπερη που είναι εκπρόσωπος του ΕΚ. Κύριε Κάσπερη, έχετε ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς ακριβώς έρχεστε εδώ ενώπιόν μας τόσο σύντομα μετά τη θέση ισχύ της Λισαβόνας. Γιατί στη Θεσμική Επιτροπή αγωνιστήκατε ως μέλος του Κοινοβουλίου για περισσότερα δικαιώματα στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πω στα δύο θέματα. Ε, στα οποία απαντήσατε ε, για τις μελλοντικές εντολές για τις διαπραγματεύσεις. Το Κοινοβούλιο, λέτε, θα πρέπει να συμμετέχει με πλήρη φωνή. Μετά όμως τη λήξη και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο δεν ε, έχει τη φωνή που θα έπρεπε. Και επίσης η κοινή εμπορική πολιτική και η κοινή εξωτερική πολιτική. Πώς διαχωρίζεται, πώς εξασφαλίζεται και πώς ε, θα εξασφαλίσετε την αυτοτέλεια και την ανεξαρτησία της εμπορικής πολιτικής για να μην θυσιάζονται αυτά σε άλλους βομούς, όπως ακούσαμε χτες, δυστυχώς, ε, σε μια άλλη ακρόαση της Επιτρόπου. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ντεχούιχτ έχει δύο λεπτά για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. το θέμα της ε, έγκαιρης εφαρμογής ε, θα το αντιμετωπίσουμε ε, με τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Κορέας. Με την συνθήκη της Λισαβόνας κάτι άλλαξε. Γίνεστε πραγματικοί συνομοθέτες και έχετε φωνή για όλες τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Η έγκαιρη εφαρμογή δεν είναι κάτι καινούριο που ξαφνικά εμφανίστηκε στι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου και μάλιστα συγκεκριμένη με την Κορέα. Είναι συνηθισμένη πρακτική του διεθνού εμπορίου. Βεβαίω καταλαβαίνω ότι η έγκαιρη εφαρμογή πριν δώσει την σύμφωνη γνώμη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Θα πρέπει στη συμφωνία πλαίσιο να το ρυθμίσουμε αυτό το θέμα. Στη συμφωνία πλαίσιο ε, με την Κορέα. Θα το συζητήσω με την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και θα δω αν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για την πρόταση για την έγκαιρη εφαρμογή. Τώρα, για την ανεξαρτησία της εμπορικής πολιτικής σε σχέση με τις άλλες πολιτικές, φυσικά η ανεξαρτησία είναι μια σχετική έννοια. Η φύση της κοινή εμπορικής πολιτικής εξασφαλίζει ότι θα κρατήσει την ανεξαρτησία της, γιατί είναι από τις λίγες αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον είσαστε και συνομοθέτες και θα πρέπει να συμφωνήσετε. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία και σε σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με αυτή την ε, υπηρεσία, αλλά δεν σημαίνει ότι θα υποταχθούμε σε αυτήν. Έχω, θα μπορούσα να σας πω και άλλα, αλλά δυστυχώς έχω μόνο δύο λεπτά. Θα έχετε την ευκαιρία, λέει ο Πρόεδρος, α, να επανέλθετε. Ο κύριος Κάσπαρη ξανά. Θα ήθελα να παραμείνω στον τομέα αυτό. Είπατε ότι η συνδίκηση της Αβώνας έχει διαμορφώσει έτσι το εξωτερικό εμπόριο, ώστε να είναι ισότιμο το Κοινοβούλιο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εσείς Πώς θα το μεταφράσετε αυτό στην πράξη, τι θα κάνετε για να πάρει σάρκα και οστά. Πώς θα διασφαλίσετε α πούμε ότι το Κοινοβούλιο σε διαδικασίες κατά του ντάμπινγκ θα συμμετέχει και στη διαβούλευση και στη λήψη των αποφάσεων. Και μια άλλη ερώτηση σε σχέση με αυτό. Ω Επίτροπος Εξωτερικού Εμπορίου ε, πηγαίνετε συχνά σε πολλέ χώρε που είναι εμπορικοί εταίροι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει συνήθεια όταν ταξιδεύουν οι υπουργοί να συνοδεύονται από βουλευτέ. Θα μπορούσατε να φανταστείτε εσεί κάτι τέτοιο, να σα συνοδεύουν ευρωβουλευτέ στι επαφέ σα ε, στο εξωτερικό, για να ε, προαχθεί και ο κοινοβουλευτικό διάλογο. Ένα λεπτό για την απάντηση, κύριε Ντεχούιτ. Για το αντι-dumping. Θα έχετε κι εσείς ε, λόγο αλλά φυσικά την απόφαση θα την πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της διαδικασίας επιτροπολογίας. Το να υπάρχουν δικαιώματα βέτο για το αντι-dumping δεν συνάδει με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά θα δείξω ανοιχτό πνεύμα για αυτό το θέμα και για το αντι-dumping θα έχω μια προσέγγιση που θα προωθεί κάποιους κανόνες που θα σέβονται τον κανονισμό αντι-dumping. Θα το συζητήσουμε ούτως ή άλλως. Τώρα, το να συνοδεύομαι από ευρωβουλευτές κάνει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω βέβαια αν έχω προϋπολογισμό για κάτι τέτοιο, γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Έπειτα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις ε, πολυμερείς διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕΑ, όπου είσαστε τμήμα της, Ευρω... της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τις διμερείς αντιπροσω... Ε, διαπραγματεύσεις. Ε, στις διμερείς ε, διαπραγματεύσεις προϋποτίθεται ότι υπάρχει και θεώρηση και ίσως είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, ο κύριος Αρίφ. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, έχετε την φήμη ότι είσαστε ε, ειλικρινείς. Εμείς εμπλεκόμαστε στην ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης Παρά τις απροθυμίες του Συμβουλίου, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε λόγο. Θα μας στηρίξετε. Ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα, στα πλαίσια του χρονικού ορίζοντα του 2020. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η θέση σας. Είμαι πεπισμένο ότι μια εμπορική πολιτική θα πρέπει να συνδεθεί με μια πραγματική βιομηχανική πολιτική που δημιουργεί και θέσει απασχόληση. Επομένω, σα θέτω το εξή ερώτημα. Ε, θα υποστηρίξετε την αεροναυπηγική α, δημόσια ε, και στην, ε, στις, ε, στον πόλεμο που υπάρχει μεταξύ των εταιριών. τι θέση θα πάρετε. Δύο λεπτά για την απάντηση. Για τη συνεργασία με την Επιτροπή σας, λέει ο κύριος Ντεχούχτ, το κοίταξα με το Γενικό Γραμματέα το θέμα και με την υπηρεσία, τις υπηρεσίες μου. Και θα ήθελα να δεσμευτώ ήδη σήμερα, μετά από τις παρατηρήσεις διαφόρων βουλευτών, θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι καταρχάς θα υπάρχει ε, μια ευρύτερη ε, και γρηγορότερη ροή πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαζί θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ε, και θα πρέπει να δούμε όμως και πώς θα χειριστούμε τα εμπιστευτικά μας έγγραφα γιατί είναι πρόβλημα και αυτό θα σας βοηθήσω για να επεξεργαστείτε το μεγάλο όγκο των πληροφοριών ε, με ad hoc ενημερώσεις. Ε, θα έχω συχνές επαφές με την Επιτροπή σας, ε, τη Γραμματεία και τα μέλη της, Επι... της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τακτικές ενημερώσεις εδώ στο Συμβούλιο, εδώ στο Κοινοβούλιο, συγγνώμη, σε περίπτωση που δεν είστε μέλη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την πρώτη και τρίτη ερώτηση, μίλησατε τόσο γρήγορα που δεν σας κατάλαβα. Ξέρω ότι έχετε λίγο χρόνο, αλλά και εγώ έχω περιορισμένη ικανότητα να απορροφήσω κάτι το οποίο διατυπώνεται τόσο γρήγορα. Δεν σας κατάλαβα, δεν είναι θέμα γλώσσας, είναι θέμα ταχύτητας. Εντάξει, μπορείτε να ε, ξαναθέσετε το ερώτημά σας λοιπόν. Για ένα λεπτό, επί ένα λεπτό. Ναι, θα το ξαναπώ λοιπόν. Έλεγα ότι μια νέα στρατηγική πρέπει να καθοδηγεί την πολιτική της Ένωσης στη όραμά της για το 2020. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σα θέση. Τέλο, έλεγα ότι μια εμπορική πολιτική πρέπει να συνδυάζεται με μια πραγματική βιομηχανική πολιτική που να δημιουργεί θέσει εργασία και η επικαιρότητα με οδηγεί να σας ρωτήσω, θα υποστηρίξατε την αερογραφική βιομηχανία, ιδιαίτερα στη διαμάχη της με τον ΠΟΕ. Uh, um, l'agenda Euh, το πρόγραμμα για το 2020 δεν μπορεί να αποτύχει γιατί ακόμη δεν έχει καν ε, διατυπωθεί. Η εμπορική πολιτική πάντως έχει κάτι, διαθέτει ένα πολύ μεγάλο ατού. Δηλαδή, είπαμε για το 2020 ότι ο κύριος στόχος είναι περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας, προσλήψεις, ε, με όλη την κοινωνική προστασία που απαιτείται βέβαια. Πάνω απ' όλα όμως ανάπτυξη. Και την ανάπτυξη, για την ανάπτυξη χρειάζεται μία σωστή εμπορική πολιτική. Υπάρχουν δύο διαμάχες. Airbus κατά Boeing και Airbus κατά Poe. η αμάχη με την Boeing προς τον Ιούνιο μάλλον θα ξεσπάσει αλλά πρέπει πρώτα πριν αποφανθούμε να έχουμε όλα τα στοιχεία γιατί η μία υπόθεση θα έχει επιπτώσει την άλλη. Είναι σχεδόν δικαστική διαδικασία και πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες της, το της προσφυγής στον ΠΟΕ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την πρώτη αυτή ερωταπάντηση. Ο κ. Δεχούς δεν εξάντλησε το χρόνο του. Λοιπόν, τώρα εκπρόσωπος των φιλελευθέρων ο κ. Καζάκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Τι φρονείτε για τις σχέσεις της εμπορικής πολιτικής με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης και τι σχέσεις θέλετε να δημιουργήσετε με την ύπατη εκπρόσωπο εξωτερικών. Θα υποστηρίξετε, θα προωθήσετε τις ιδιαιτερότητες, θα προασπίσετε τις ιδιαιτερότητες που έχει η εμπορική πολιτική και πώς θα πετύχετε το στόχο να μην υποκύψει σε συγκεκριμένα συμφέροντα η πολιτική αυτή. Δεύτερον, οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις που θα οργανώσετε με εκπροσώπους ε, ε, οργανώσεων εμπόρων. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά για την απάντηση από τον κύριο Ντεχούχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εμπορική πολιτική είναι τμήμα της εξωτερικής. Αλλά επίσης έχει και ιδιαιτερότητες. Όπως είχα ήδη πει στον κύριο Κάσπαρη, είναι αποκλειστική δικαιοδοσία. Η Κομισιόν έχει τις περισσότερες δικαιοδοσίες για το θέμα αυτό γιατί εκείνη διαπραγματεύεται τις εμπορικές συμφωνίες και μάλιστα θα έχει και περισσότερες δικαιοδοσίες από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Άρα τα εργαλεία που διαθέτουμε uh, για τη δράση μας διεθνώς είναι ακόμη περισσότερα. Επομένως οι σχέσεις με την υπάτη εκπρόσωπο είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και για τα εμπορικά θέματα. Παραδείγματο χάρη θέματα αντι-dumping. Φαντάζομαι ότι παρά τους κανόνες που ήδη υπάρχουν, τους τεχνικούς κανόνες θα χρειαστούν και πολιτικές συζητήσεις και θα γίνουν, θα γίνουν. Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα. Η πάτη εκπρόσωπος είναι εξάλλου η προηγούμενη εμπορική επίτροπος, άρα ξέρει πολύ καλά τα εμπορικά θέματα. Όσο για την παρουσία σε διεθνείς διασκέψεις και στον ΠΟΕ, είναι και αυτό ένα πραγματικό θέμα. Αλλά στην Επιτροπή 1.33 είναι πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί πρέπει να υπάρξει συμφωνία με το Συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί ή συζητήθηκε στη Συμφωνία Πλαίσιο αλλά διαφέρει βέβαια από το ερώτημα προηγουμένως που θέσατε για τις διεθνείς εμπορικές διασκέψεις. Ο κύριος Καζάρ συμπληρωματική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να τύχει κάποια ερμηνεία, ε, δηλαδή να δούμε με ποιου κανόνες θα εφαρμοστεί η συνεργασία των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα όμως να μα πείτε, να μας επιβεβαιώσετε ότι είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα συμμετέχει σε όλες τις διαπραγματεύσεις και ότι η παρουσία του, την παρουσία του μπορείτε να την εγγυηθείτε στην Επιτροπή 1.33. Θα μας δίνετε τις πληροφορίες τις ίδιες που δίνεται και στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Μονόλεπτη απάντηση. Για τα έγγραφα της Επιτροπής κανένα πρόβλημα θα έχετε ακριβώς τα ίδια με το Συμβούλιο και ταυτόχρονα. Και έχει και αυτό τη σημασία του. Όχι μόνο ποια έγγραφα αλλά και πότε. Όσο για τα έγγραφα άλλων ομάδων που θα συμμετέχουν, χωρών, συμβουλίου κτλ. Αυτό είναι άλλο θέμα, άλλο πράγμα. Θα έχετε επίσης τα αποτελέσματα των μελετών που αναλαμβάνουμε, το σχεδιασμό τους. Θα είμαι όσο το δυνατό πιο ανοιχτό με το Κοινοβούλιο. Εξάλλου ήμουν και εγώ για 15 χρόνια Ευρωβουλευτής και είμαι υπέρ της αύξησης των δικαιοδοσιών του. Δεν άλλαξε η στάση μου, μόνο η θέση μου άλλαξε. Τώρα που είμαι από την άλλη πλευρά της τραπέζης μαζί με τις χώρες μέλη, το Συμβούλιο και τους άλλους επιτρόπους, μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μου. Και τώρα ο πρόσωπος των Πρασίνων, ο κύριος Ζαντού. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, η στρατηγική που είχε καθοριστεί, η εμπορική στρατηγική, είχε καθοριστεί πριν να ξεσπάσουν οι κρίσεις και οι κλιματολογικές αλλαγές. Εμείς θεωρούμε ότι η στρατηγική λοιπόν αυτή τελικά περιορίζεται στα αυστηρά εμπορικά τεχνικά θέματα Θεωρείτε λοιπόν ότι τα υπόλοιπα όπως οι κλιματολογικές αλλαγές είναι λεπτομέρειες που δεν έχετε το χρόνο να ασχοληθείτε με αυτές ή θα τα κάνετε, θα τα στήσετε αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής. Ευχαριστώ. Μόνο λεπτή απάντηση. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπεύθυνο για την εμπορική πολιτική. Οι υπόλοιπες πτυχές που αναφέρατε εξαρτώνται και ε, ασχολούνται με αυτές άλλοι επίτροποι. Και επειδή η Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, θα ήθελα να τονίσω ότι η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να ασκηθεί εν κενό. Έχει επιπτώσεις στο δημοσιονομικό σύστημα, στο χρηματοπιστωτικό, στις υπηρεσίες, Είδαμε τι έγινε με τη χρηματοπιστωτική κρίση. Υπάρχει το κλιματολογικό θέμα. Είδαμε βέβαια ότι στην Κοπενχάγη τα αποτελέσματα ήταν πολύ μέτρια. Η εμπορική λοιπόν πολιτική θα μπορούσε ίσως να συμβάλλει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Διότι, διότι η χρηματοδότηση της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών από τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι κάτι που μπορεί να προκύψει από την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων. Είναι λοιπόν ζωτικό και ουσιώδες να έχουμε μια σφαιρική αντιμετώπιση, ολιστική. Συχνά συμβαίνει αυτό σε πολιτικά θέματα γιατί δεν μπορεί κανείς να απομονώσει τα προβλήματα το ένα από το άλλο. Πάντοτε είναι χρήσιμη μια σφαιρική προσέγγιση, αλλά επίσης δεν πρέπει να γνωρούμε ότι οι αρμόδιοι για τα θέματα που θίξατε είναι άλλοι, όχι εγώ. Και πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνεργασία. Εγώ πάντως σφαιρικά θα το βλέπω, σφαιρικά, σφαιρικά. Ευχαριστώ μονόλεπτη συμπληρωματική. Οι δικαιοδοσίε σας αφορούν τις εξαιρέσεις που χορηγούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, παραδείγματος χάρη σε συμφωνία με την Νότια Κορέα, όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, ο φόρος προσαρμογής στα σύνορα. Τέλος, υπήρξαν τεθαραλέως, ως προς τη δημοκρατία, δημοκρατία δηλαδή του Κονγκό θα δείξετε το ίδιο θάρρος και για την Κολομβία. Μονόλεπτη ανταπάντηση. Α, κοιτάξτε. Το θέμα της Κολομβίας θα επανέλθει σίγουρα. Δεν μου αρκεί ένα λεπτό για να απαντήσω και για τα δύο θέματα που θίξατε. Λοιπόν, για τα σύνορα, εγώ είμαι κατά. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή λύση είναι κάτι που θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, το έχουμε δει ήδη και στο παρελθόν. Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι να καταλήξουμε σε εμπορικό πόλεμο. Είναι φανερό ότι πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα για την εμπορική πολιτική από όσα συμβαίνουν και σχετικά με τις κλιματολογικές αλλαγές και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επίσης μια πιο στεναρή πολιτική προσέγγιση που να μην διαφωνεί με τους κανόνες της αγοράς. Ευχαριστούμε. Και τώρα εκπρόσωπος των συντηρητικών, Ζάχερ Σαράντιο. εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μητρική μου, την τσεχική. Και θα κάνω μια ερώτηση για τη Ρωσία. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι επίκειται νέα συμφωνία με τη Ρωσία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε αυτή τη σχέση, στρατηγική εταιρική σχέση, θεωρείτε ότι είναι ένα νέο εργαλείο, η συμφωνία που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε ε, τους εμπορικούς φραγμούς, μη τελωνιακούς εννοώ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά αυτή τη διάσταση της κατάργησης των διακρίσεων και της πρόσβασης στους ενεργειακούς πόρους, όπως είναι το φυσικό αέριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια επίσης. Δύο λεπτά για την απάντηση, κύριε Ντεχόχτ. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Η ενεργειακή ασφάλεια βεβαίως είναι ένα θέμα πάρα πολύ κρίσιμο και το εμπόριο έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει καθώς και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ας πούμε για τις συμφωνίες ελευθέρω εμπορίου αυτό το καιρό κάνουμε διαπραγματεύσεις και με την Ουκρανία και είναι αρμόδια ε, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου γι' αυτό. Σε όλες όμως τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και σε άλλες διαπραγματεύσεις ε, λαμβάνεται αυτό δεόντως υπόψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που να γίνονται σεβαστές σε ένα πλαίσιο τέτοιο συμφωνιών. Και εδώ μιλώ και για ένα μηχανισμό διακανονισμού των διαφορών που είναι από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ε, των ε, συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Το άλλο ερώτημά σας για τους μη τελωνιακούς εμπορικούς φραγμούς. Προσωπικά είμαι επιπισμένο ότι αυτό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την εμπορική μα πολιτική τα ερχόμενα έτη. Ακόμα περισσότερο από τι ίδιε συμφωνίε εμπορικέ. Γιατί όταν έχουμε εμπορικέ συμφωνίε και στον ΠΟΕ καταργούμε του τελωνιακού φραγμού, και μετά βλέπουμε να αναδύονται μαζικά ε, μη τελωνιακοί φραγμοί. Το είδαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια δεκαετία αγωνιστήκαμε για να ε, καταργήσουμε στην Ευρώπη φραγμούς άλλους πλην των τελωνιακών. Όλο και περισσότερο λοιπόν θα δούμε τέτοια εμπόδια και ο καθένας θα ε, αναπτύξει και κάποια ειδικότητα. Αλλά τουλάχιστον τα επόμενα έτη σας λέγω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να λύνεται περισσότερο διμερός και πολυμερός και λιγότερο σε επίπεδο ΠΟΕ, διότι εκεί δεν έχουμε ακόμα τα σωστά εργαλεία και τις σωστές συμφωνίες που χρειαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και ε, θα το χειριστώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Συμπληρωματική ερώτηση για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω εγώ ε, με την ερώτηση αυτή για τη Ρωσία. Εσείς υποστηρίζετε την ένταξη της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, λαμβανωμένου υπόψη επίσης και του θέματος των σχέσεών της με τη Λευκορωσία και το Καζαχστάν. Και θα πρέπει να υπάρξει και συμφωνία σύνδεσης με τη Λευκορωσία και το Καζαχστάν θα πρέπει να μπουν στη γειτονία αυτά τα κράτη. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό για να απαντήσετε, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Βεβαίως και υποστηρίζω την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Αλλά από τους Ρώσους εξαρτάται. Έχουν συνάψει αυτή τη τελωνιακή σχέση με τη Λευκορωσία και το Καζαχστάν και παρόλο που δήλωσε ο πρόεδρος Μετβέντεφ ε, στη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο, αν δεν απατώμε, ότι θα προσπαθήσουν να μπουν στον ΠΟΕ συντομότερο, πρέπει να δούμε στην πράξη τι σημαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, Πού δίδουν μεγαλύτερο βάρος και προτεραιότητα στη Τελωνιακή Ένωση με άλλες χώρες ή στον ΠΟΕ, γιατί αυτό έχει σημασία και για τους δασμούς. Έχουν αυξηθεί. Και βλέπετε ότι η Ρωσία σήμερα δρά αντίθετα ε, με κάποιες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και υποχρεώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με την ένταξή του στον ΠΟΕ. Βεβαίως ε, είναι προσωρινά τα μέτρα αυτά, αλλά δούμε τι θα σημάνουν στην πράξη. Όλα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα. Τώρα για τις συμφωνίες ελευθέρω αν μου δώσετε περισσότερο χρόνο, Πρόεδρε, μπορεί και να απαντήσω. Σε άλλη απάντηση, μελλοντική να επανέλθετε. Τώρα δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της ομάδας ερωτικής αριστεράς, γοέ, τον κύριο Σόλτς. Κύριε Υποψήφιο επίτροπε πρέπει να σας λέω. <laughs> Στις προτεραιότητες σας μιλήσατε για το γύρο της Δόχα και για τον ΠΟΕ και για την Ατζέντα 2020. Έτσι δηλώνεται ως προτεραιότητα. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω την εξής συμπληρωματική ερώτηση. Ποια είναι η δική σας ανάλυση για την αποτυχία του γύρου της Ντόχα μέχρι στιγμής. Ποια είναι τα αίτια. Και δεδομένη της αποτυχίας, εσείς θέλετε να συνεχίσετε να διαπραγματεύεστε με τον παλιό τρόπο ή μήπως θεωρείτε ότι η παλιά εντολή του 2010 που ήταν δεινόσαυρος για μένα και προέρχεται από το έτος 2001. Μήπως θα πρέπει λέγω να προσαρμοστεί στις σημερινές πραγματικότητες ε, της οικονομίας της παγκόσμιας, ιδιαίτερα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Thank you. minutes for reply. If you wish, you could come back to the other question if you have the time. Um, Παρακαλώ, απαντήστε και αν θέλετε και στην προηγούμενη ερώτηση αν έχετε χρόνο. Για τα αίτια της αποτυχίας δεν θα μιλούσα για αποτυχία γιατί συμφωνούμε στο 90% των θεμάτων. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει αυτές και αν δεν γίνει αυτό το 2010 τότε το 2011. Είμαι αισιόδοξο, επαναλαμβάνω. Και γι' αυτό σας είπα ότι είναι και υπαριθμόν ένα προτεραιότητα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Τώρα τι θα γίνει μετά θα δούμε. Και για την εντολή, όχι, να μην αλλάξουμε την εντολή. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει τώρα η εντολή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι μόνο χρονοβόρο και περιπλέκει τα πράγματα. Και βέβαια δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα με το γύρο της Δόχα, αλλά υπάρχει και χρόνος μετά. Αυτό που θα προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε και θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω να ολοκληρωθεί η συμφωνία το συντομότερο. Ξέρω ότι γίνονται και άλλα ερωτήματα μήπως πρέπει να αλλάξουμε το μηχανισμό λήψη αποφάσεων, μα ε, δεν είναι ρεαλιστικά αυτά. Για να ολοκληρωθεί ο γύρος της Δόχα και να προχωρήσουμε στη συνένεση, αυτή είναι η μόνη δυνατότητα σε πολυμερές επίπεδο. Και αν τελικά αποτύχει, θα συμφωνήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα και η Ινδία. Δηλαδή ακόμα και αν υπάρχει η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία θα έχουμε και το θέμα της ανησυχηρίας του ΒΕΤΟ. Το θέμα δεν είναι δηλαδή να λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, πλειοψηφικά, αλλά έχουμε βασικές διαφορές απόψεων για θέματα σημαντικά και ε, ε, το πιο σημαντικό είναι η γεωργία σε αυτό. Συμπληρωματική ερώτηση, ο κύριος Σόλτς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι, αλλά δεν θεωρείτε παρόλα αυτά ότι και σε σχέση με τα όσα ρώτησε ο κύριο ε, Ζαντό για το κλίμα, για την επισητιστική κρίση, την πείνα, τη φτώχεια στον κόσμο, δεν χρειάζεται ακριβώς αυτή η αλλαγή νοοτροπία στον ΠΟΕ και δεν θα είχε νόημα. Ξέρω εγώ, πέρα από την προσωπική σας άποψη για την τόχα που μας την αναφέρατε, δεν θα μπορούσατε να προβληματιστείτε γενικότερα για το πώς μπορεί ε, ο ΠΟΕ ο ίδιος να μεταρρυθμιστεί για να ασχολείται με τέτοια θέματα διαφορετικά, για το κλίμα, για το βληθισμό, για τους ανθρώπους. Είπατε ότι είναι το καλύτερο μοντέλο συνεργασία αυτό. Μήπω χρειάζεται όμω αλλαγή στην νοοτροπία Και τότε να έχουμε ένα νέο μηχανισμό κοινοβουλευτική συνέλευση. Δηλαδή, να συγκεντρώνονται άνθρωποι από όλες τις χώρες και να προσπαθήσουν να ε, αναδιαμορφώσουν το εμπόριο για ε, σημαντική αναπτυξιακή συνεργασία με διαφάνεια. ένα λεπτό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο γύρος της Ντόχα που δημιουργήθηκε ως αναπτυξιακός γύρος να έχει και αποτελέσματα, να δώσει αποτελέσματα σε επίπεδο ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό για τις αντισώμενες χώρες, για τη σχέση των ε, χωρών του Βορρά και του Νότου, αλλά και τη σχέση των χωρών του Νότου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε στεναροί υποστηριχτές ε, της ε, διάστασης ανάπτυξης. Και αυτό προϋποθέτει ότι θα δούμε και τα θέματα κλιματικής αλλαγής και το πώς το εμπόριο μπορεί να συνεισφέρει. Γιατί η χρηματοδότηση θα πρέπει από κάπου να προκύψει. Και κυρίως από την οικονομική ανάπτυξη ε, στις αντισόμενες χώρες. Πέρα από τα δημόσια κονδύλια. Τώρα, για το αν και κατά πόσο ο ΠΟΕ θα πρέπει να έχει μια ευρύτερη ατζέντα και για το αν θα πρέπει να αντιμετωπίσει και προβλήματα κλιματικών αλλαγών. Η εμπορική διάσταση θα πρέπει να συζητείται επίσης και στον ΠΟΕ και γίνεται ούτως ή άλλως αυτό, αλλά για μια διεθνή οργάνωση είναι σημαντικό να κρατήσει την εστίασή της να μην διασπαθίζεται σε, πολλές, σε πολλούς στόχους. Ο ΠΟΕ είναι, μια, είναι μια οργάνωση που ε, ποιοτικά ε, είναι ανώτερο σε επίπεδο οργάνωσης από τον ΟΗΕ. Ε, θα σταματήσουμε εδώ κύριε Ντεχούχτ. Τώρα οι Ευρωπαίοι Ελεύθεροι Δημοκράτες. Ο κύριος Ντάρτμουθ. Κύριε υποψήφιε επιτροπή. τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικές οικονομίες, διαφορετικής δομής, διαφορετικά χαρακτηριστικά στις οικονομίες τους και διαφορετικές εμπορικές πολιτικές. Παρ' όλα αυτά, η μόνη εκπροσώπηση που τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό και το, και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, έχουν στον ΠΟΕ είναι μέσω του Επιτρόπου εμπορικής πολιτικής. Εσείς ως τέτοιος ε, επίτροπος πώς θα μπορέσετε να προωθήσετε πλήρω και ισότιμα τα εμπορικά συμφέροντα όλων των 27 κρατών μελών και κυρίως μια και έχετε μια πλήρη πολιτική ατζέντα που την αναφέρατε δύο φορές ε, στις παρατηρήσεις σας. Πώς θα μπορέσετε όλα αυτά τα, πράγματα δηλαδή να τα, παντρέψετε μεταξύ τους. Δύο λεπτά για την απάντηση τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ε, εξασφαλίζουν ότι μπορεί να καταλήξει σε μια κοινή θέση και να την υπερασπιστεί αποτελεσματικά στα διεθνή φόρουμ. Την παρατήρηση που κάνετε για την εμπορική πολιτική μπορεί να την κάνετε για οποιαδήποτε πολιτική. Φυσικά είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας. Είμαστε 27 και έχουμε αναβαθμίσει τους μηχανισμούς λήψη αποφάσεων στη συνθήκη της Λισαβόνας. Το κάναμε και για το εμπόριο. Το Κοινοβούλιο θα εμπλακεί πλήρως. Φυσικά δεν υπάρχουν μόνο πολιτικές διαφορές στο Κοινοβούλιο, αλλά και εθνικές διαφορές. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βοηθάει για να ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές. Ε, νομίζω ότι εκεί έγκυται η διαφορά μας. Έχουμε διαφορε... διαφορετικές απόψεις εσείς και εγώ. Αλλά γι' αυτό είσαστε... Ε, υπάρχει το κοινοβούλιο, εσείς έχετε την άποψή σας ε, και την εκφράζετε, αλλά εγώ ως Επίτροπος εκφράζω όχι την προσωπική μου γνώμη, την... αλλά την άποψη του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια το θέμα είναι τεράστιο. Ε, έχει και πολλές πολιτικές αποχρώσεις. Ε, θεωρώ ότι είναι καλύτερο που έχουμε ένα ε, επίτροπο για θέματα εμπορικής πολιτικής. Φανταστείτε να υπήρχαν περισσότεροι για αυτή τη δουλειά, δεν θα υπήρχε συμφωνία. Ε, ένα λεπτό για την συμπληρωματική ερώτηση. Ε, μου δώσατε απάντηση σε δύο λεφτά σε μια τόσο περίπλοκη ερώτηση. Είμαι Βρετανός βουλευτής. Το 1973 μπήκαμε στην τότε κοινή αγορά και είχαμε τότε ένα ε, μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα με τις χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, έκτοτε έχουμε ένα τεράστιο και αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα. Ίσως τελικά καλύτερα θα ήταν να είχαμε τη δική μας εκπροσώπηση, εφόσον έχουμε έτσι τα πράγματα. Α, και παρεμπιπτόντος. Σας παρακαλώ, Πρόεδρε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω και μία άλλη ερώτηση να μας πείτε κάτι για τα πολιτικά σας, ε, πιστεύω, τις πολιτικές, τους πολιτικούς σας στόχους. Γιατί στις γραπτές σας απαντήσεις το αναφέρατε αυτό σε τρία-τέσσερα σημεία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε και άλλα στοιχεία. Ίσως είναι καλή ιδέα το ότι η πρώτη σας ερώτηση ε, συζητείται κιόλας ε, στο Westminster, στη Βρετανία εγώ δεν έχω άποψη γι' αυτό. Ε, το εμπόριο αναπτύχθηκε πάρα πολύ στη δεκαετία του 70 και του 80. Ε, επομένως, πολιτικά είναι αυτά τα θέματα, δεν μπορώ να τα συζητήσω εγώ. Ε, τώρα, για την πολιτική μου ατζέντα. Είμαι πεπισμένος ότι η εμπορική μας πολιτική εξυπηρετείται καλύτερα από μια πιο ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουμε ανεξάρτητοι, να κρατήσουμε την ιδιαιτερότητά μας, γιατί αλλιώς θα γίνουν πιο δυσχερείς οι διαπραγματεύσεις. Προφανώς η πολιτική διάσταση ε, έχει το πρώτο, τον πρώτο λόγο, την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με την εμπορική διάσταση. Και η εμπορική πολιτική δεν βασίζεται μόνο σε οικονομική βάση. Ε, γι' αυτό είναι πολύ καλή ιδέα το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, έχουν αυτή την εμπλοκή για τα, τις αρμοδιότητες του είπα του εκπροσώπου. Και τώρα προχωρούμε σε μια δεύτερη δέσμη ερωτήσεων. Ερωτήσεις από τις επιτροπές που ασχολούνται με την εμπορική πολιτική. Η ΔΕΒΕ, δηλαδή η Επιτροπή Ανάπτυξης και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η κυρία Ζολή ε, είναι πρόεδρος της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Έχει το λόγο. Τέσσερα λεπτά συνολικά. Ένα λεπτό η αρχική ερώτηση, ένα λεπτό η απάντηση, ένα λεπτό η συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό η συμπληρωματική απάντηση. Κυρία Σολή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ντεχούχτ να μας δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς θα εξασφαλίσει ότι οι νέες εμπορικές συμφωνίες συνάδου με το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας, που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας στις πολιτικές που εφαρμόζει και που μπορεί να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για να ερμηνευτεί αυτό το άρθρο, είσαστε ε, διατεθειμένος να καταφύγετε μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ένα λεπτό για την απάντηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι αυτή τη στιγμή επίτροπος ε, ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή. Όχι για πολύ ακόμα. Αλλά δεν ξεχνάω αυτή τη θέση. Και θα, ήθελα ε, το αποτέλεσμα του γύρου της Ντόχα να δώσει και αντιξιακά αποτελέσματα. Είναι σημαντικό για τις αντισώμενες χώρες. Είμαι πεπισμένος πραγματικά ότι αν οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν γίνουν τμήμα της ε, παγκόσμιας οικονομίας, δεν έχουν πραγματικό μέλλον. Για την Αφρική, ας πούμε. Αν αναπτυχθεί το εμπόριο, θα βοηθηθεί η Αφρική. Ε, δεν θα πρέπει οι σχέσεις μόνο βορρά-νότου ε, να αναπτυχθούν, αλλά και σχέσεις νότου-νότου. Οι εμπορικές συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις αναπτυξιακές ε, ε, πτυχές υπόψη. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθεί πραγματικά η Αφρική. Συμπληρωματική ερώτηση. Παρακαλώ για ένα λεπτό η κυρία Ζολή. Δεν έχω συμπληρωματική ερώτηση. Από την Επιτροπή Εξωτερικών, ο κύριος Πρόβερα. On my left. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντεχούχτα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ε, αποτελείται ε, κατά το 90% από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα βοηθήσουν για να καταπολεμηθεί ο αθέμητος ανταγωνισμός μέσα σε, μια, σε ένα οικονομικό παγκόσμιο πλαίσιο όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι δύσκολος. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα εμπορικής άμυνας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενδυναμωθεί. Μετά από τις δυσκολίες που είχαμε με τις ΕΠΑ για να εναρμονίσουμε την ε, εμπορική νομοθεσία και με την Κίνα για την καταπολέμηση της ε, απομίμησης και για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, η Κομισιόν τι σκοπεύει να κάνει για να αναπτύξει πιο ισορροπημένες οικονομικές σχέσεις ε, και εμπορικές σχέσεις μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτών των εταίρων, της Κίνας δηλαδή και των ΗΠΑ. Ένα λεπτό για την απάντηση του κ. Ντεχούχτ. Ε, Κύριε Προβέρα, σωστά είπατε ότι πολλές από τις ευρωπαϊκές ε, οικονομίες βασίζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βεβαίως οι μικρομεσαίες είναι πολύ πιο ευάλωτες σε φραγμούς μη δασμολογικούς ε, από ότι κάποιες πολυεθνικές εταιρείες. Και βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Και όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα σε όλες τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που κάνουμε με τρίτες χώρες ή με ε, ομάδες τρίτων χωρών. Σε ό,τι αφορά τα συστήματα, συστήματα προστασίας του εμπορίου, σας είπα εισαγωγικά ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν, αλλά αυτά να τα κάνουμε μετά το πέρας ε, του γύρου της ε, Ντόχα, της ολοκλήρωσης δηλαδή των διαπραγματεύσεων και βάσει των εμπειριών μας πλέον. Στη συνέχεια, αν δείτε τον όγκο του εμπορίου, ε, που αναφέρεται είναι μόλις το 2% και με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες 98%. Εγώ είμαι πάντα υπέρ των κανόνων και μιας προσέγγισης συγκροτημένης και χωρίς να μπαίνουμε σε πάρα πολιτικά ε, θέματα. Ευχαριστώ. Συμπροματική ερώτηση για ένα λεπτό. Για τις διμερείς εμπορικές ε, συμφωνίες, ε, ποιες στρατηγικές θα ενεργοποιήσει η Κομισιόν ούτως ώστε να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις με σημαντικές ε, ομάδες, γεωγραφικές ομάδες του η ομίλους του πλανήτη, όπως το Μερκοσούρ και το ΑΖΕΑΝ. Εμείς είμαστε υπέρ της περιφερειακής προσέγγισης. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα, γιατί όχι, δεν είναι πάντα όλες οι χώρες της περιοχής στο ίδιο επίπεδο, όπως την ε, ΑΖΕΑΝ παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό και η Κομισιόν πρότεινε και το Συμβούλιο δέχτηκε αυτή την πρόταση. Πρότεινε λοιπόν να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις διαπραγματεύσεις και να ξεκινήσουμε διμερείς διαπραγματεύσεις, κυρίως με τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη μέσα σε μια όμω ε, περιφερειακή πολιτική προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν, οι υπόλοιπε χώρε. Τώρα, με το Mercosur, ε, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Οι συζητήσει σταμάτησαν το 2004. Είμαστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε. Ε, υπό τον όρο όμως ότι και οι εταίροι μας συμφωνούν. Καλό θα ήταν να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά χρειάζονται και οι δύο. Και οι δύο πρέπει να συμφωνούν για κάτι τέτοιο. Και τώρα περνάμε σε, στον τρίτο γύρο των ερωτήσεων. Με ερωτήσει από τα μέλη της Επιτροπής. Ξεκινάμε με την κυρία Σάιφη από το ΕΛΚΑ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθουμε στα μέτρα αντι-dumping. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και νομίζω ότι θα πρέπει να επαγρυπνήσουμε και σε αυτήν εδώ την κοινοβουλευτική θητεία. Ξέρετε ότι η βιομηχανία μας χρειάζεται μέτρα αντι-dumping που να είναι αποτελεσματικά για να καταπολεμήσουμε την, τον αθέμητο ανταγωνισμό και στις ε, αρχικές παρατηρήσεις σας μας είπατε ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιες πρακτικές αθέμητου εμπορίου. Συμφωνώ απόλυτα επίσης και με αυτό που είπατε ότι το ελεύθερο εμπόριο δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αφέλεια. Μα είπατε ότι αυτά τα μέτρα αντι-dumping θα τα βελτιώσετε. Δώστε μα σας παρακαλώ περισσότερες ε, λεπτομέρειες. Θα έχουμε ανοιχτά τα μάτια, γιατί ο Πίτερ Μέντελσον, ο προκάτοχός σας, ε, ενώ έλεγε ότι θα τι βελτιώσει, αυτές τις, ε, αυτά τα μέτρα αντι-dumping, στην πραγματικότητα τα αποδυνάμωσε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω περισσότερε λεπτομέρειε. Ένα λεπτό για την απάντηση. Ευχαριστώ. Ήδη έχω απαντήσει σε κάποιο βαθμό σε αυτό το ερώτημα. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε το τέλος του γύρου της Ντόχα υπό τον όρο ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Θα προωθήσω αυτά τα μέτρα, το είπα και, στα, και στη δήλωσή μου. Αν φοβάστε ότι θα είμαι πιο χαλαρός, πιο ανεκτικός, όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική πολιτική αντι-dumping. Που να είναι αξιόπιστη και που οι εταίροι μας ξέρουν πολύ καλά τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Να είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό για να λειτουργεί και ως αντικίνητρο. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ατού μας όταν χρειάζεται. Πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε και το κουράγιο να δράσουμε όταν χρειάζεται. Είμαι πεπισμένο ότι σε ορισμένε περιπτώσει χρειάζονται τέτοια μέτρα αντι-dumping. Σε ορισμένε περιπτώσει. Αλλά δεν θα πρέπει να υπερεκτιμήσουμε ε, τη σημασία αυτών των μέτρων. Ε, ένα λεπτό για την ε, συμπληρωματική ερώτηση. Δεν μας δώσατε ουσιαστικές λεπτομέρειες, αλλά θα μας τις δώσετε φαντάζομαι στο μέλλον. Θα διατηρήσετε την ανεξαρτησία των αρχών που είναι επιφορτισμένες με τις έρευνες. θα εξασφαλίσετε ότι οι βασικές αρχές του κανονισμού αντι-dumping θα παραμείνουν αλόβητες και δεσμεύεστε να διαβουλευτείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Ευχαριστώ. Οι υπηρεσίες που διενεργούν αυτές τις έρευνες είναι ανεξάρτητες, ε, δουλεύουν με αξιόπιστο τρόπο και οποιοδήποτε διαδικασία αντι-dumping ξεκινάει με μια τέτοια επαγγελματική έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσουν και να γίνουν αυτές οι έρευνες με, με τρόπο ανεξάρτητο. Επίσης θα πρέπει να κρατήσουμε ε, και όλα τα πλεονεκτήματα, όλα τα του, του κανονισμού αντι-dumping και της πολιτής αντι-dumping αλλά ενδεχομένως ε, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Αλλά γενικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια πολιτική αντιτάμπη στο σημερινό εμπορικό κλίμα. Ε, στο μέλλον ίσως θα πρέπει να προσαρμόσουμε αυτή την πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει πιο χαλαρή καθόλου. Ε. Και τώρα δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κύριο Ντέιβιτ Μάρτιν. Ένα λεπτό για ερώτηση. Ευχαριστώ. Κάρελ, σε ξέρω από παλιά είσαι ειλικρινής και ισχυρός πολιτικός, αλλά σήμερα απογοητεύτηκα γιατί ε, λες, έχω και τις, ε, συνήθως λες ε, τις προσωπικές απόψεις και όχι του κολεγίου των επιτρόπων. Όταν έρχεσαι εδώ, θέλουμε να ακούμε τις δικές σου απόψεις και συγκεκριμένα σήμερα. Τη δική σου γνώμη θέλω και όχι του κολεγίου των επιτρόπων για την συνοχή και τη συνέχεια. Ξέρεις ότι ως Επίτροπος Ανάπτυξης ότι ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για την καταπολέμηση του AIDS και άλλων νόσων στον κόσμο. Και μετά κάνουμε διάφορες πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες ε, στα TRIPS, ε, TRIPS ε, Plus όπως λέγονται στον ΠΟΕ. Και ξέρω ότι κάποιοι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά την αντίθετη γνώμη του Κοινοβουλίου, συνεχίζουν αυτή τη τακτική και προωθούν τέτοια θέματα TRIPS Plus στις συμφωνίες. Απάντηση. Καταρχάς, Νομίζω ότι κατά 99% η προσωπική μου άποψη στο θέμα αυτό το χαρτοφυλακείο μου ταυτίζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπόλοιπο 1% επιτρέψτε μου σήμερα να το κρατήσω για τον εαυτό μου. Πέρα από όλα αυτά όμως πιστεύω στεναρά ότι κάθε άνθρωπος έχει ε, θεμελιώδης δικαίωμα πρόσβηση στα φάρμακα. Το θέμα δεν είναι εύκολο. Έχει να κάνει με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι δική μας πολιτική και είναι η διαφύλαξη των δικαιωμάτων αυτών. Και πιστεύω ότι το πράττουμε και στην τελωνιακή μας πολιτική, παρόλο που υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά αν τη μελετήσετε θα δείτε ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν να φτάνουν τα φάρμακα στον προορισμό τους. Γνωρίζω ότι γίνεται μια συζήτηση που λέει αν θα πρέπει να έχουμε διατάξεις τύπου TRIPS plus ε, ορισμένες ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Δεν είμαι κατά ανάγκη αντίθετος με αυτό το μέτρο, αλλά νομίζω υπάρχει δυνατότητα να το δούμε και διαφορετικά. Να υπάρχουν τέτοιε διατάξει για συγκεκριμένα προϊόντα και συγκεκριμένα αίτια και από την άλλη αυτό να αντισταθμίζεται από παράλληλες εισαγωγέ, Φερρυπίν. Μάλιστα. Μονόλεπτη συμπληρωματική. Παρόλα αυτά προτίθεστε να αναθεωρήσετε την οδηγία για τους δασμούς 1383 ιδιαίτερα ως προς την Ινδία γιατί αυτή έχει μεγάλη σχέση με τα φάρμακα η Ινδία παράγει πολλά φάρμακα και οι φραγμοί δεν βλάπτουν μόνο την ίδια αλλά και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες η συμφωνία με την Ινδία ακόμη την χάνει διαπραγμάτευσης. Θα παρακολουθήσω από πολύ κοντά να φροντίσω, θα φροντίσω να μην παρεμποδιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία φτηνών φαρμάκων χωρίς copyright. Δεν αποκλείω μία εξαίρεση τύπου TRIPS-SYN η γενικότερη ιδέα είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα αυτά και πράγματι θα ζητήσω αναθεώρηση της οδηγίας που αναφέρατε. Αλλά θα χρειαστεί βέβαια κάποιος χρόνος. Χρειάζονται πάντως σίγουρα προσαρμογές για να αποφευχθούν αυτά που έγιναν στην Ολλανδία πρόσφατα. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Κουίς Χάρντα του ΕΛΚ για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε θερμότατα στα Ολλανδικά, κύριε υποψήφιε ε, Επίτροπε για το Εμπόριο και ελπίζω να έχουμε και καλή συνεργασία. Νομίζω ότι είμαι η μόνη Γερμανίδα φλαμανδικής καταγωγής εδώ στην Επιτροπή μας και επιστρέφω στα γερμανικά. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπατε για τη Ρωσία. Θεωρείται και το σημείωσα ότι είναι πολύ σημαντικό κράτος η Ρωσία για τις εμπορικές μας σχέσεις. Γεγονός είναι αυτό άλλωστε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης βλέπετε ότι ανάλογα με την προέλευση κάθε βουλευτού διαφέρει η άποψή του με το τι πρέπει να κάνουμε με τη Ρωσία. Είπατε ότι δεν ξέρετε καν αν θέλει η ίδια η Ρωσία να μπει στον ΠΟΕ. Γι' αυτό ε, κάνω και την εξής ερώτηση. Πώς φαντάζεστε τώρα το μέλλον και τις εμπορικές μας σχέσεις με τη Ρωσία. Πώς μπορούμε να τις αναπτύξουμε είτε είναι μέλος των ΠΟΕ είτε δεν είναι. Πώς θέλετε αυτά όλα να τα κάνετε σε συνεργασία με την Επίτροπο και ε, την εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Ε, το βλέπετε μόνο ρεαλιστικά, τεχνοκρατικά ή και πιο πολιτικά. Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί απάντηση σε αυτή την ερώτηση σε 60 δευτερόλεπτα. Πιστεύω όμως ότι έχουμε θεμελιώδες ε, ενδιαφέρον και συμφέρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε καλή σχέσεις με τη Ρωσία. Είτε αυτές είναι πολιτικές είτε είναι οικονομικές. Αυτό νομίζω διαφυλάσσεται ως εξή. Να έχουμε συμβατικές υποχρεώσεις. Γι' αυτό και η συμφωνία που αυτό τον καιρό διαπραγματευόμαστε με τη Ρωσία είναι τόσο σημαντική. Το εμπορικό κεφάλαιο να είναι πολύ καλά ανεπτυγμένο. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι καλό το γεγονό ότι η Ρωσία ε, θα πρέπει να ενταχθεί στον ΠΟΕ το συντομότερο, γιατί και εκεί υπάρχουν σημαντικέ υποχρεώσει και δεσμεύεται να τη στείλει η Ρωσία. Αλλά και πολιτικά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί είναι γειτονέ μα και θα παραμείνουν γειτονέ μα. Τι να κάνουμε. Οπότε έχουμε κάθε συμφέρον να έχουμε τέτοιες σχέσει μαζί τους. Από την άλλη, δεν μπορώ παρά να παραδεχθώ ότι αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουμε προβλήματα. Παράδειγμα στο εμπόριο, διότι έχουν ε, βάλει ε, μονομερός πολλούς δασμούς και μπορούν αυτό το καιρό ακόμα να το κάνουν, παρόλο που υποσχέθηκαν το αντίθετο στη συμφωνία μας, ε, στη σχέση με τον ΠΟΕ. Πολλά λοιπόν από τα θέματα αυτά θα αντιμετωπίζονται πιο εύκολα ή θα αντιμετωπίζονταν αν ήταν πιο σαφείς συμβατικές υποχρεώσεις και για τα δύο μέρη. Μόνο 50 δευτερόλεπτα συμπληρωματική ερώτηση, γιατί στην πρώτη ερώτηση ξεπεράσετε κατά πολύ το χρόνο σας. Και πάλι έχει σχέση με τη Ρωσία η ερώτησή μου, όχι όμως μόνο με τη Ρωσία. Είναι πολύ σημαντικό για την ενεργειακή μας ασφάλεια και τον ανεφοδιασμό να έχουμε αξιόπιστους εταίρους και να μπορούμε να υπολογίζουμε σε, στις παραδόσεις ε, της ενέργειας αυτής και στον ανεφοδιασμό και με άλλους εταίρους, όχι μόνο με τη Ρωσία, αλλά την Ουκρανία, το Ιράν, το Ιράκ κλπ. Πώς βλέπετε συγκεκριμένα εσείς αυτή τη συνεργασία και τι θέλετε να κάνετε έτσι ώστε ο ρόλος του Επιτρόπου Αρμοδίου για θέματα εμπορίου και της Επιτροπής μας να μην ε, εξαφανιστεί κάπου σε αυτή την περίπλοκη συνεργασία. Έχω και άλλη ερώτηση όμως τώρα, πάρα πολύ σύντομη. Η συνάδελφός μου, κυρία Σαϊφή, σας ρώτησε αν προτίθεστε να ε, συμπεριλαμβάνετε το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις ε, κατά του ντάμπινγκ. Ε, θέλετε ναι ή όχι, είναι απλή απάντηση. Για οφνές τα Ολλανδικά. σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις κατά του ντάμπινγκ, τις διαπραγματεύσεις αυτές, αυτές. Αυτό είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει τις διαπραγματεύσεις αυτές. Είμαι πρόθυμος να το συζητήσω μαζί σας αν θέλετε και να ακούσω προσεκτικά τις προτάσεις σας. Οι διαπραγματεύσει οι ίδιες όμως είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφήστε που πιστεύω ότι είναι καλύτερα έτσι. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την προμήθεια ε, και την ασφάλεια ανεφοδιασμού ενεργειακού εννοώ, εγώ δεν φοβούμαι ότι τελικά η ανεξαρτησία της εμπορικής μας πολιτικής ε, θα αποδυναμωθεί, ας πούμε. Αντίθετα, πιστεύω ότι ακριβώς επειδή αναπτύσσουμε περισσότερο τις εξωτερικές μας οικονομικές ε, σχέσεις και πολιτικά και εμπορικά βγαίνουμε ενισχυμένοι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεργαστώ με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αλλά δεν είμαι τμήμα αυτής της υπηρεσίας. Ε, ε, εγώ αγαπώ πάρα πολύ την ανεξαρτησία και είναι καλό που είμαστε ανεξάρτητοι. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι εκεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σούστα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, από την οποία δεν έχουμε ακόμη εξέλθει, απαιτεί μία σειρά νομοθετικά μέτρα που θα συνοδεύουν την οικονομία για να βγει από την κρίση και τη βιομηχανία επίσης. Τι πρόταση έχετε να, κάνετε για την πρόταση κανονισμού για το εμπορικό σήμα για να προστατευτούν οι, εμπο, οι καταναλωτές. Ε, πριν από λίγε εβδομάδε πήρε θέση με μεγάλη πλειοψηφία το Κοινοβούλιο υπέρ. Και τι προτάσει έχετε για να καταπολεμηθεί ε, η απομίμηση των προϊόντων ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, παγκόσμια. Έπειτα, για τη συμφωνία με την Κορέα. Θα πρέπει να δούμε τι επίπτωση θα έχει στην πραγματική οικονομία και να μην το δούμε το θέμα μόνο ακαδημαϊκά. Ε, υπάρχει επίσης ο κίνδυνος ε, να ε, πλήξει πολλούς παραγωγικούς τομείς στην Ιταλία αλλά και στην Ευρώπη. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό. Ένα λεπτό για την απάντηση κύριε Ντεχούχτ. Ξέρετε ότι υπάρχει διαφορά απόψεων για την πρόταση αυτή ε, για το σήμα. Το Κοινοβούλιο είναι υπέρ και το Συμβούλιο είναι κατά. Θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε μια πρόταση η προκάτοχός μα, η κάθε Άστον, έκανε κάποιες προτάσεις τον Οκτώβριο και ελπίζω αυτές οι νέες προτάσεις να διευκολύνουν την διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Τώρα, οι απομιμήσεις προϊόντων, τα ψευδεπίγραφα προϊόντα. Ξέρω πολύ καλά ότι οι υποστηρικτές της οδηγίας, και μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να αποφασιστεί με συναπόφαση, λένε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις απομιμήσεις, ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια καλή συμφωνία για την καταπολέμηση της, των απομιμήσεων. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ό,τι μπορούμε ε, και να έχουμε αποτελέσματα απτά και στα πλαίσια του ΠΟΕ για αυτό το θέμα. Μία διευκρίνηση για το θέμα της Κορέας. Νομίζω ότι για αυτή τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Κορέα θα μπορούσατε να πείτε δύο λόγια παραπάνω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Κορέα. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που θα πρέπει να τους ε, συζητήσουμε, παραδείγματο χάρη τα αυτοκίνητα, αλλά σε ό,τι αφορά τα κλωστοϊφαντουργικά, η Συμφωνία ε, ούτως ή άλλως οι εμπορικές ροές ε, είναι πολύ μικρές σε αυτόν τον τομέα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας. Ε, η συμφωνία αυτή ε, έχει κάποιες βασικές διατάξεις και κάποια μέτρα διαφύλαξης που μπορούν να δρομολογηθούν μετά από μια περίοδο τεσσάρων χρόνων. Μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα το συντομότερο δυνατόν αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα, πραγματικά εγείρονται προβλήματα στον τομέα της ε, βιομηχανίας. Από το ΕΛΚ, ο κ. Γουίνκλερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να παραθέσω κάτι που είπατε το πρωί. Είπατε ότι για να υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη, το εμπόριο ε, μπορεί να παίξει το ρόλο της ατμομηχανής. Εγώ είμαι Ρουμάνος και σημείωσα με ικανοποίηση αυτή την δήλωση. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας για τη σημασία και το ρόλο της Συμφωνίας ΣΕΦΤΑ ε, του 2006. Είναι πολύτιμο εργαλείο για να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών ε, Βαλκανίων. Η συμφωνία αυτή ΣΕΦΤΑ του 2006 είναι μια προπαρασκευαστική προσπάθεια ε, για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ε, προκειμένου να εφαρμόσουν την κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θεωρείται γενικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Συμφωνείτε με τη δική μου άποψη. Η ΣΕΦΤΑ είναι τμήμα της προενταξιακής διαδικασίας. Να μην ξεχνάμε ότι ένα νέο κράτος μέλος δεν είναι εύκολο να χωνέψει μονομιάς όλο το κοινοτικό κεκτημένο. Γιατί έχουμε πολύ ανεπτυγμένες τις οικονομικές διαστά, ε, πτυχές και γι' αυτό ακριβώς ε, βάσει συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου ε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις χώρες να καταργήσουν ε, τα, τους μη τελωνιακούς δασμούς. Είναι ένας ε, μηχανισμός ολοκλήρωσης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυτικών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ο πολιτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν όχι το συντομότερο δυνατό μόνο, αλλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολιτικά αλλά και οικονομικά. και είναι πολύ σημαντικό και για τα ιστορικά και ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Συμπληρωματική ερώτηση. Στην ανακοίνωσή σας προς το στο Κοινοβούλιο είπατε ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα ε, συμπληρώνεται από αποτελεσματικές διμερείς ε, συμφωνίες. Ε, σε αυτό το πλαίσιο, τι σχέση έχει τέτοιες συμφωνίες με την Ουκρανία ή, με τη Μολδαβία, η οποία ήταν τμήμα του, της συμφωνίας ΣΕΦΤΑ του 2006. Ε, η ερώτησή μου είναι η εξή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εμπόριο, το εμπόριο ως εργαλείο για να προσεγγίσετε αυτές τις χώρες ε, για να αποκτήσουν μια ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν θα δεσμευτώ στην, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας. Θα πρέπει να το αφήσουμε κατά μέρο αυτό το θέμα. Καταρχάς θα πρέπει να γίνει τμήμα του ΕΟΧΑ, Με την ευρύτερη έννοια. Για τη Μολδαβία επίσης υπάρχουν και πολιτικά προβλήματα, όπως ξέρετε, τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Επομένως πρέπει να έχουμε μια βαθμία προσέγγιση. Ε, στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας έχουμε αυτή τη βαθμία προσέγγιση ε, που είναι και προσαρμοσμένη στις, ε, στην κάθε χώρα. Και μέσα αυτή την προσέγγιση που είναι εστιασμένη στην κάθε χώρα, η ΣΕΦΤΑ είναι πολύτιμο εργαλείο. Θέλουμε να την εντάξουμε τη Μολδαβία, αλλά το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό μόνο. Καταλαβαίνω ότι ο ίσως Ρουμάνος ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα, αλλά υπάρχουν και πολιτικές, πολιτικά προβλήματα, πολιτικές ευαισθησίες σε σχέση με τη Μολδαβία. Ο κύριος Ρινάλντι, εκπρόσωπος του Άλντε, των Φιλελεύθερων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, πολλές συγκεκριμένες ερωτήσεις ακούστηκαν. Εγώ τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω ε, για αυτό που είπατε στον κύριο Ρίφ Είπατε ότι ο στόχος του διεθνούς εμπορίου είναι η ανάπτυξη, η απασχόληση ε, με σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ε, και ότι την ανάπτυξη θα πρέπει να τη βρούμε συχνά και αλλού. Εγώ είμαι νέο μέλος Συχνά όταν συζητάμε με την Κομισιόν για κάποια δεδομένα, παραδείγματο χάρη η συμφωνία για την Κορέα, με βάση κάποιε πληροφορίε που έχουμε, μπορεί να οδηγήσει σε πολλέ απώλειε ε, θέσεων εργασία. Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα τα τελευταία πέντε χρόνια τριπλασιάστηκε. Όταν συζητάμε με του συνομιλητέ ΑΚΕ, λένε ότι η συμφωνίες, ναι μεν αυξάνουν το εμπόριο με τις χώρες τους, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα σε κοινωνικό επίπεδο και στον παραγωγικό του τομέα. Θα ήθελα να μου πείτε, ποια είναι, κατά, κατά την αποψή σας, οι παράμετροι επιτυχίας μιας εμπορικής πολιτικής. Εάν η αύξηση, είναι μήπως ας πούμε η αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών ή είναι κάποια κριτήρια αξιολόγησης ε, της πραγματικής οικονομίας. Uh, uh, Πράγματι το έλλειμμα έχει αυξηθεί. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Όπως στην την Ασία στο σύνολό της, θα έπρεπε να πούμε ότι τα θέματα των ελλημάτων αλλάζουν από χώρα σε χώρα. Εκεί. Ο στόχος μας δεν είναι η αύξηση του εμπορίου κάθε αυτού, αλλά το γεφύρωμα των χασμάτων και η εξισορρόπηση. Δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμια οικονομία βέβαια χωρίς εμπόριο και για να υπάρξει διεθνές εμπόριο χρειάζονται διεθνείς κανόνες. Αυτό είναι η δουλειά μου. Δεν είναι απλώς η προώθηση του εμπορίου. Αυτό είναι θέμα των χωρών μελών. Μερικές φορές και των περιφερειών τους. Εγώ θέλω να καθοριστεί το πολιτικό και νομικό πλαίσιο που να καθιστά δυνατή την σωστή άσκηση του εμπορίου με προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών διεθνώς και παγκοσμίως. Πραγματική ερώτηση. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, όταν ε, ταξιδεύετε, ε, θα ήθελα να πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ασία. Ε, υπάρχουν κάποια διασκεδαστικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για προϊόντα μεγάλης κατανάλωσης, τα οποία είναι απομιμήσεις και πουλούνται, λες και είχαν παραχθεί όπως νόμιμα λοιπά, όπως πουλούνται τα νόμιμα προϊόντα στην Ευρώπη. Προτείνεται την επέκταση του άρθρου 23 των TRIPS που σήμερα περιορίζεται στα αλκοολούχα ποτά και σε άλλα προϊόντα που έχουν ευρωπαϊκή γεωγραφική προέλευση απλό μέτρο, το οποίο θα μπορούσε όμως σε διεθνή φόρουμ να εξασφαλίσει πραγματική προστασία αυτών των γεωγραφικών ενδείξεων. Ένα λεπτό για την απάντηση. Έχω ταξιδέψει και εγώ, έχω δει τα πράγματα, ήμουν υπουργό εξωτερικών, έχω δει ορισμένες αγορές και χώρες τρίτες αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί κανείς να επεκτείνει το 23 όπως ζητάτε παραδείγματος χάρη και για την παραγωγή των αγαθών, ορισμένων αγαθών τουλάχιστον. Χρειάζεται συμφωνία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για όλα αυτά για περιορισμό του εύρους που θα είναι απόφευκτος άμα γίνουν αυτές οι προτάσεις αλλά απ' την άλλη για το TRIPS δεν νομίζω ότι μπορούν να συγκριθούν τα ποτά με τα παπούτσια για να το πω έτσι. Και τώρα το λόγο κύριε Στάτσνη και πάλι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, στις 15 Οκτωβρίου, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Η Κάθριν Νάστον, προκάτοχό σα, υπέγραψε συμφωνία ελευθέρω εμπορίου με την Νότιο Κορέα. Και τώρα η συμφωνία αυτή αναμένει ε, την εκύρωσή της από τα κράτη-μέλη και το παρόν κοινοβούλιο. Έχω και ειδική ερώτηση. Γνωρίζετε ότι οι υποχωρήσεις που δίνονται στη ε, Κορέα ε, για να μην αναγράφεται η προέλευση ενός προϊόντος θα είναι εις βάρος των Ευρωπαίων κατασκευαστών που έρχονται να ανταγωνιστούν τα κορεατικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα υπάρχουν ίσοι κανόνες παιχνιδιού στην ευρωπαϊκή αγορά και θα ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο. Ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι είναι πολύ έμφαδες και λεπτό αυτό το θέμα. Προσπάθησα να καταλάβω ακριβώς περί τίνος πρόκειται και να συνειδητοποιήσω και τις επιπτώσεις και τις συνέπειες. Και με απλούς υπολογισμούς καταλήγω στο εξή συμπέρασμα. Ένα αυτοκίνητο που κοστίζει 10.000 ε, ευρώ θα έχει αντίκτυπο ε, της τάξης των 100 ευρώ. Εντάξει, Ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να συζητούμε τα θέματα σε βάθος. Από την άλλη, αυτή η υποχώρηση και η κατάργηση duty drawback, αυτό είναι μια διεθνής πρακτική ε, αναγνωρισμένη και την ε, επικαλείται και η Ευρώπη. Δεν εμφανίστηκε από το πουθενά αυτό με την Κορέα ξαφνικά. Εάν υπάρχουν όμως προβλήματα μπορούμε να αντιδράσουμε. Υπάρχει ειδικό μηχανισμός που έχει προβλεφθεί και μπορούμε να το περιορίσουμε στο 5% ενώ αυτό τον καιρό είναι γύρω στο 8%. Και περιορίζεται λοιπόν και αντίδραση μπορούμε να έχουμε με ασφαλιστικές δικλείδες και μέτρα μπορούμε να ε, λάβουμε. Σε περίπτωση που έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία σας αναφέρετε, υπάρχουν μηχανισμοί και δυνατότητες δράσης και αντίδρασης. Ας κρίνουμε όμως με βάση τις επιδόσεις στη συμφωνία και θα δούμε στο μέλλον τι θα προκύψει. Συμπληρωματική ερώτηση. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός κάπως. Και είπατε και στην εισαγωγή σας ότι είναι καλή η συμφωνία. Το καλός για μένα σημαίνει μια μέτρια συμφωνία. Ε, και κάθε φορά που έχουμε μέτριες συμφωνίες ε, είναι δυσαρεστημένοι οι ενδιαφερόμενοι. Εσείς μπορεί να θεωρείτε ότι ε, δεν θα έχουμε κατασκευή βιομηχανικών και παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων στην Ευρώπη, αλλά θα τα εισάγουμε. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ κακό για τις θέσεις απασχόλησης. Δεν τηρήσετε το χρόνο σας στην πρώτη απάντηση, αυστηρά ένα λεπτό. Τι θα πει μέτρια. Το καλός για μένα σημαίνει καλός. Δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή ο όρος μέτριος. Η καλή συμφωνία είναι καλή. Η λέξη σημαίνει αυτό που σημαίνουν. Λοιπόν, θα δούμε την εφαρμογή τη συμφωνίας, πώς θα πάει. Έχουμε ασφαλιστικές δικλίδες. Σας είπα, είμαστε πρόθυμοι να σας διαβιβάσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε για να υποστηρίξουμε τη θέση μας ότι πραγματικά είναι επωφελής η συμφωνία αυτή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι και για την κατασκευαστική βιομηχανία στην Ευρώπη θα είναι καλή. Και δεν είναι πρόβλημα στην ουσία. Έχουμε, επαναλαμβάνω, ε, ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση εμφάνισης ανισορροπιών. Αν δείτε αυτά τα βιομηχανικά προϊόντα, η Νότια Κορέα δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ασία. Έχουμε και άλλα προβλήματα εκεί που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και σίγουρα δεν είναι η Κορέα, γιατί το βιωτικό του επίπεδο είναι πολύ υψηλότερο. Ε, σε όλα τα επίπεδα γενικά είναι πιο ανεπτυγμένοι και αναλαμβάνουν και υποχρεώσεις οποίες ε, σέβονται στα πλαίσια των συνθηκών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, ή τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πώς να το πω, ε, δεν είναι το υπαριθμό ένα πρόβλημα στην Ασία από πλευρά βιομηχανικών προϊόντων. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες τώρα. Η κυρία Μουνή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις σχέσεις ε, με τη Λατινική Αμερική ε, και την κοινότητα των Άνδεων υπάρχει μια κόπωση και έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το αναφέρει. Και τελικά ορισμένα από τα μέλη του Συμφώνου των Άνδεων έχουν αρχίσει διμερείς ε, διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ αναφέρομαι στο Περού και την Κολομβία. Για την Κολομβία υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο σέβεται τα συνδικαλιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Ορισμένοι θεωρούν ότι η παραβίαση είναι σοβαρή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνει συμφωνία με την Κολομβία και κάποιοι άλλοι λένε ότι η κατάσταση βελτιώνεται αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, έχουμε ε, τυπικές σχέσεις και σύσφυξη των δεσμών μας με τη χώρα αυτή για να μπορέσουμε ακριβώς να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά. Uh, Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια τεχνική αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μεταβεί στη Λίμα ε, για ε, περαιτέρω διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. Υποθέτω ότι δεν θα καταλήξουμε σε απόφαση δεν θα ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, διότι παραμένουν ζητήματα προς συζήτηση, αλλά ε, επαναλαμβάνω είναι σε τεχνικό επίπεδο οι επαφές, όχι σε πολιτικό. Εν πάση περιπτώσει. Θα μονογράψουμε συμφωνία με την Κολομβία μόνο εφόσον γίνει βαθύτατη συζήτηση για το θέμα αυτό. τεχνικές συζητήσεις είναι αυτές και μόνο και δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα έχουμε μονογραφή της συμφωνίας. Μόνο μετά από βαθιά πολιτική συζήτηση θα προχωρήσουμε. Πραγματική ερώτηση. Ε, ναι. Για τον ΠΟΕ θέλω να ρωτήσω και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Θέλουν να βγουν απ' έξω ε, τα ποτά και τα, τα και οι ίνοι που έχουν ε, γεωγραφική ονομασία προέλευσης. Εσείς ε, πώς το βλέπετε αυτό, πώς το εκτιμάτε. discussion uh, Η συζήτηση στα πλαίσια του ΠΟΕ συνεχίζεται για τις λεγόμενες γεωγραφικές ενδείξεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση το βλέπουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άλλωστε. Ξανά και ξανά επανέρχεται συνεχώς το θέμα. Και θα αποσκοπήσουμε σε μια φιλόδοξη συμφωνία και στον ΠΟΕ για το θέμα αυτό. Το συζητούμε και σε διμερείς διαπραγματεύσεις και σε περιφερειακές αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο φιλοδοξούμε να έχουμε πραγματικά μια τέτοια συμφωνία. Και τώρα ήρθε η ώρα των πρασίνων. Η κυρία Κάρολάιν Λούκας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για την επιρροή που έχουν οι μεγάλες εταιρείε στην ευρωπαϊκή πολιτική. Στη γραπτή απάντηση στα ερωτήματά μας λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία, ανεξάρτητο ρόλο τη ε, υπηρεσία σα και συμπεραίνεται ότι η ανεξαρτησία είναι κάτι το τελείως ζωτικό για να προστατευτούμε από επενδεδημένα συμφέροντα. Μου αρέσουν αυτά τα λόγια και θα προσέχουμε ιδιαίτερα να δούμε αν θα τα εφαρμόσετε. Ιδιαίτερα ως προς τη στρατηγική της Λισαβόνας που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βαρόσος Μερικοί όμως έχουμε την εντύπωση ότι μετά από την εμπειρία των προκατόχων σας και ορισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων που απέδειξαν με προσφυγές ότι παρά τις επανειλημμένες επαφές και διασκέψεις έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει επιρροή των εταιριών στην στρατηγική, θα ήθελα να μου πείτε πώς θα έλξει ο χρόνος. μα είναι θέμα προσωπικής ακαιρεότητος. Εγώ είμαι υπέρ της πλήρους διαφάνειας και για τις υπηρεσίες μας και για τους λομπιίστες και λομπιίστριες. Ξέρετε ότι είναι πια αναπόφευκτη η παρουσία τους. Έχω συναντηθεί με τον πρόεδρο του Business Europe που είναι φυσικά από τους συνομιλητές μας φυσικότατα και θα τον ξανασυναντήσω και είμαι διατεθειμένος να κάνω διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών uh, και όπως έγινε με τον Επίτροπο Λαμή πριν από 10 χρόνια. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώς παίζεται στις διαπραγματεύσεις και αυτό μπορούμε να το μάθουμε μόνο αν συναντήσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους και θα το κάνουμε ίσες αποστάσεις. Συμπληρωματική. Ναι, ίσες αποστάσεις, αλλά το θέμα δεν είναι η πρόσβαση των λομπιστών, αλλά το ποσοστό τους, η σημασία τους Στην προηγούμενη καριέρα σας είχατε δημιουργήσει ένα βελγικό σώμα διαβούλευσης με μεγάλους επιχειρηματίες, αλλά δεν συμπληρώσατε και με προσώπους της κοινωνίας των πολιτών και συνδικαλιστών. Μπορείτε να μας υποσχεθείτε ότι ως Επίτροπος θα λάβετε υπόψη σας και αυτούς τους ενδιαφερόμενους για να είναι πιο ισορροπημένη η εκπροσώπηση. Είχα πει και προηγουμένως ότι δεν είναι ίδιος ο ρόλος μιας χώρας μέλου και της Ένωσης στο σύνολό της. Μια χώρα μέλος πρέπει να προωθήσει τα εμπορικά της συμφέροντα. Εγώ το εμπορικό συμβούλιο που αναφέρατε, το επιχειρηματικό συμβούλιο μάλλον, το δημιούργησα για να προωθηθεί η πώληση, η εξαγωγή ορισμένων βελικών προϊόντων σε τρίτες χώρες. αλλά και ως υπουργό ε- Εξωτερικών επίσης είχα κάνει διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των, της κοινωνίας των πολιτών εξαμηνιές για γενικότερα θέματα, με διαβουλεύσεις για γενικότερα θέματα εξωτερικής πολιτικής του Βελιγίου. Και πάντοτε είχα την πόρτα μου ανοιχτή αν ήθελαν να προσφύγουν σε μένα. Και το ίδιο θα κάνω και στη νέα μου θέση. Ευχαριστούμε. Τελείωσε ο πρώτος γύρος. Και τώρα αρχίζει ο δεύτερος ε, των προσκεκλημένων επιτροπών. Η κυρία Στρίφλερ. Στρίφλερ, Μιχαήλα Στρίφλερ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα που επετέχθη συμφωνία στον ΠΟΕ για τη διένεξη μεταξύ ΙΠΑ και Ένωσης για τις Βανάνες, τι μέτρα θα λάβετε ώστε οι χώρες ακένα να είναι σε θέση να συνεχίσουν να παράγουν βανάνες με ανταγωνιστικό τρόπο στη διεθνή αγορά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν στο κοινωνικό δάμπινγκ. Καταρχήν χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί υπήρξε συμφωνία επί των βανανών. Γιατί αν θέλουμε να λήξει όντως ο γύρο της Δόχας χρειάζεται και συμφωνία για τις μπανάνες. Πολύ σημαντική συμφωνία. Πολύ σημαντική. Όσο και οι μπανάνες οι ίδιες. Γιατί Πρόκειται για μείωση κατά περίπου 80% γενικότερα των δασμών, ενώ για τις μανάνες μόνο 35%. Αυτά λόγω της πρώιμης ε, συγκομιδής. Θα χρειαστούν 200 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των τοπικών παραγωγών βανάνης για τις χώρες ΑΚΕ αλλά και για τους Ευρωπαίους παραγωγούς βανάνης. Υπάρχει τέτοια παραγωγή. Και υπάρχει το λεγόμενο Green Box που πληρώνει άμεσες στηρίξεις για τους παραγωγούς βανάνης. Ο εκπρόσωπος της ΕΠΕΞ Μιλτσέα. Πάσχος Μιλτσέα. Ευχαριστώ πολύ. Με τη θέση του υπάτου εκπροσώπου θελήσαμε να δώσουμε μια μεγαλύτερη συνοχή στη συντονισμό των δραστηριοτήτων εξωτερικών δράσεων και σχέσεων. Άρα, όπως το είπατε ήδη, πρέπει να συνεργάζεστε και ως εμπορικός επίτροπος με την υπάτη αυτή εκπρόσωπο. Αλλά απ' την άλλη, τι φρονείτε για τις συμφωνίες συνεργασίας και τις εταιρικές συμφωνίες σε σχέση με τις καθαρές εμπορικές συμφωνίες. Τι σχέση υπάρχει μεταξύ των δύο. Ευχαριστώ. Η διαφορά είναι ότι μία συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών έχει δίνει προτεραιότητα στο εμπόριο και άρα στον εμπορικό επίτροπο. Ενώ στην εταιρική συμφωνία η πάτη εκπρόσωπος έχει το προβάδισμα. Αυτή είναι η διαφορά. Η δε απόφαση του κατά πόσον η συμφωνία είναι ελευθέρου εμπορίου ή εταιρική για, και για άλλα δηλαδή θέματα, όχι μόνο εμπορικά. Υπάρχουν πολλά αρχικά, όπως ξέρετε, που τα περιγράφουν όλα αυτά. Είναι πολιτική απόφαση και λαμβάνεται από το Συμβούλιο προτάση της Κομισιόν. Συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις σύναψης εταιρικών συμφωνιών με τη Ρωσία και για το εμπορικό του τμήμα διασφαλίζουμε ή θα διασφαλίσουμε σοβαρότατο ρόλο στις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι πολιτική καταρχάς η απόφαση αυτή του χαρακτήρα της συμφωνίας. Οι εταιρικέ πάντως δεν είναι μόνο εμπορικές, αλλά αφορούν και άλλα θέματα. Πολύ καλό το ερώτημά όμως, μου άρεσε ιδιαίτερα συμπληρωματική. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχω συμπληρωματική, επειδή σας άρεσε. Λοιπόν, και τώρα συνεχίζεται ο δεύτερος γύρος, αλλά για τα μέλη των επιτροπών. Ο κύριος Ζάραντιλ. Ζάραντιλ. Τώρα θα είμαι πιο τεχνικός. Ακούσαμε πολλά για τη Συμφωνία της Λισαβόνας. Δεν είμαστε όλοι μας ικανοποιημένοι από αυτά που ακούσαμε, αλλά υπάρχει η Συμφωνία της Λισαβόνας και δημιουργεί και αυτή την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων που μπορεί μερικές φορές να κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα αντί να τα διευκολύνει. Ρωτώ λοιπόν κύριε Ντεχούχτ, πώς θα συντονίσετε τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου με την εξωτερική υπηρεσία ώστε να εφαρμοστεί καλύτερα η εξωτερική στρατηγική. Παραδείγματο χάρη. Οι ομάδες τοπικών αγορών θα συνεργάζονται ή όχι με τις γενικότερες εξωτερικές υπηρεσίες. το εμπόριο δεν είναι τμήμα της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων, είναι άλλο. Γιατί εκεί υπάρχουν αποκλειστικές δικαιοδοσίες, αλλά απ' την άλλη είναι πολύτιμο να υπάρχει συνεργασία με την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων που θα υπάρχει και στις Βρυξέλλες και σε τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα δε στις τρίτες αυτές χώρες, και μερικές από αυτές τουλάχιστον, έχουμε εμπορικές αντιπροσωπείες και συνεργαζόμαστε με αυτές χωρίς να είμαστε τμήμα της. Αυτή είναι υπεύθυνη στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου το οποίο όμως δεν πρέπει να είναι τμήμα της εξωτερικής υπηρεσίας, αλλά απλώς να συνεργάζεται. Δεν το φοβάμαι όμως, δεν το φοβάμαι καθόλου, διότι στο εξωτερικό της Ένωσης υπάρχουν οι εκπροσωπήσεις που γνωρίζετε πρεσβείες και τα λοιπά και βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη πολύ καλή συνεργασία και εθνικά άρα το ίδιο θα γίνει και ενωσιακά με την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου δηλαδή και την Εξωτερική Υπηρεσία. Πληρωματική για την απελευθέρωση των αγορών. Ο κύριος Μαρόσο μας είπε πολλά για την απελευθέρωση των αγορών. Σκοπεύετε λοιπόν να συνεργαστείτε ενεργά με τον κύριο Μαρόσο στα σχέδια του αυτά παραδείγματος χάρη για να ταυτίσετε τα τμήματα του κοινοτικού κεκτημένου που δεν είναι και τόσο φιλικά προς το εμπόριο. Αυτά θα καταργηθούν ή θα... Α, ο πρόεδρος. Είπα ότι πρέπει να σχετίζεται η δεύτερη ερώτηση με την πρώτη, αλλά τέλος πάντων. Δεν με πειράζει, ας απαντήσω. Ο κύριος Μπαρόσο είναι το αφεντικό μου, επομένως δεν πρέπει απλώς να τον βοηθάω, είμαι και υποχρεωμένος. Την ενωσιακή νομοθεσία μπορεί κανείς να την ερμηνεύσει με διάφορους τρόπους. Όντως όσοι ασχολούνται με το εμπόριο λένε ότι υπάρχουν μερικά μέτρα που είναι εχθρικά προς αυτό, αλλά το ίδιο ή κάτι ανάλογο μπορούν να πούν όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη, με τα διαρθρωτικά ταμεία, με τα φορολογικά κλπ. Αλλά η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι συμβιβασμός, το ξέρετε αυτό. Αν έχετε πιο συγκεκριμένη ερώτηση για συγκεκριμένα μέτρα μπορώ να τα κρίνω, αλλά γενικά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει εχθρική προς το εμπόριο νομοθεσία στην Ένωση. Ο κύριος Χίντς της Γκουε. Στο ερωτηματολόγιο σας είχατε κάποια πιεστική συμπεριφορά θέλετε να προχωρήσετε πιο γρήγορα και πιο μπροστά για τις ελεύθερες ε, συμφωνίες εμπορικές, οικονομικές κτλ. Μα υπάρχουν ε, οι πολυεθνικές που είναι ευρωπαϊκές κατακλείζουν τις αγορές της αναπτυσσόμενες χώρες, καταστρέφουν ε, εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης όπως ε, στην προτινόμενη ευρωμεσογειακή συνεργασία και γονατίζουν ε, τις χώρες αυτές. Εσείς θέλετε λέτε, να προωθήσετε όλα αυτά, έτσι, να προωθήσετε τα γυμνά συμφέροντα των πολυεθνικών. Δεν υπάρχει εδώ σύγκρουση συμφερόντων των υπερκερδών των ευρωπαϊκών πολυεθνικών με τους φτωχούς λαούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα Ίσως να διαφέρουμε λίγο στην προσέγγιση μας για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας πω τα εξή δύο. Πρώτο, δεν πιστεύω ότι μια χώρα μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν αναπτύξει την οικονομία της. Και δεν μπορεί να αναπτύξει την οικονομία της αν δεν αναπτύξει το εμπόριό της. Όταν δεν έχεις εμπόριο, για παράδειγμα στα γεωργικά προϊόντα, έχουμε ε, τη ε, γεωργία μόνο της επιβίωσης. Ε, μόνο όταν υπάρχει εμπόριο προωθείται και η εμπορική παραγωγή της γεωργίας. Γιατί ελεύθερη αγορά τώρα, το λέω και ξεκάθαρα άλλωστε τη γραπτή μου δήλωση. Στόχος της εμπορικής μας πολιτικής είναι μεταξύ άλλων να προωθούμε και τις αξίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την κλιματική αλλαγή, για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και θα είναι αναπόσπαστο ε, τμήμα αυτό της προσέγγισης μου της εμπορικής πολιτικής. Συμπληρωματική ερώτηση του κυρίου Χιγκίνης το εμπόριο μπορεί να είναι και ε, ε, βάση για την ανθρώπινη ε, αλληλεγγύη ή μπορεί να είναι βάση για μια στρεβλή σχέση όπως ισχυρίζομαι εγώ. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα λέτε ότι μόνο μετά από πολιτική συζήτηση θα προχωρείτε σε υπογραφή τη συμφωνία πούμε, με την Κολομβία. Μα οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ε, κάποιες γνωστές μάλιστα έχουν ε, ξεκάθαρα στιγματίσει και την κυβέρνησή τους και 43 παρακαλώ πολυεθνικές μεταξύ αυτών και ευρωπαϊκές για το ρόλο τους στα συνδικάτα. 49 συνδικαλιστές ε, δολοφονήθηκαν το 2008 και πάνω από 40 το 2009 και ποιος υποφελείται μεγάλες επιχειρήσεις και ευρωπαϊκές από αυτή την καταστολή κατά των συνδικάτων. Εσείς τι θα κάνετε για να διερευνήσετε αυτή την κατάσταση πριν καν σας περάσει από το μυαλό, πριν διανοηθείτε να υπογράψετε συμφωνία με την Κολομβία. Αυτό που είπα είναι ότι δεν πρόκειται να μονογράψουμε τη συμφωνία πριν ε, από τη βαθιά πολιτική συζήτηση. Πώς γίνεται μια εμπορική συμφωνία. Πρώτα έχουμε μια διαπραγμάτευση, μετά έχουμε μονογραφή, initialing και μετά υπογραφή. Εγώ είπα ότι η πολιτική συζήτηση θα γίνει πριν τη μονογραφή. Ε, θα το μελετήσουμε λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά. Στη συνέχεια, στο κείμενο της διαπραγμάτευσης μέχρι τώρα έχουμε διάταξη και ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που μπορούν να λαμβάνουν τη μέτρα και θα ληφθούν σε περίπτωση παραβίασης. Είναι όμως μια δέσμευση από πλευρά μου ότι θα υπάρξει πολιτική συζήτηση και θα δω πώς θα ε, συνεννοηθώ με τους ομολόγους μου πριν καν μονογράψουμε τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλντερ τώρα, από την ομάδα ε, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας είπα ότι γνωρίζω τον Επίτροπο. Έχουμε ε, και ε, ένα παρελθόν μαζί, όχι πάντα ειρηνικό, αλλά γενικά. Ε, στα Δυτικά Βαλκάνια βλέπουμε καρτέλ που κυριαρχούν στην αγορά, κάποιοι μεγιστάνες βλέπουμε και μάλιστα σε χώρες που προσβλέπουν στην ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ορθώνουν εμπορικά εμπόδια. Εσείς πώς θα τα αντιμετωπίζετε αυτά και είναι και επίγον το θέμα. Αν γίνεται, ε, δείτε τι γίνεται με το εισόδημα του πληθυσμού ε, τις υπηρεσίες, ε, τα τρόφιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης και ξέρω ότι είστε ευαίσθητο στα θέματα αυτά. Ε, πώς θα καταρρίψουμε αυτούς τους φραγμούς. Μιλάτε για μεγιστάνες, τα Είναι ένα πρόβλημα αυτό και τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια. Είναι γεγονός. Αλλά αυτοί οι μεγιστάνες θα μικρύνουν όταν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα περιοριστεί αυτό το γεγονός. Και αυτό ε, το αντίθετο είναι η πολιτική ανταγωνισμού. Δεν είναι δικό μου χαρτοφυλάκιο. Να ρωτήσετε τον συνάδελφό μου αν θέλετε, αλλά είμαι πεπισμένος ότι ακριβώς η ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει να καταργηθούν κάποια ιστορικά μονοπόλια και να έχουμε οικονομία της αγοράς και καλύτερα προϊόντα και σε φθηνότερες τιμές. Συμπληρωματική ερώτηση. Την επίκεια σας, Πρόεδρε, επικαλούμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι και είναι και επίγον. Ρώτησα και τη Βαρόνια ε, Άσον, την προκάτοχό σας, πέρυσι, τι γίνεται με τις ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου ε, για την καταπολέμηση ε, της παιδικής εργασίας σε θέματα έτσι εμπορίου και στις διεθνείς διαπραγματεύσει. Ο υποψήφιος ο επίτροπος μπορεί να μας πει περίπου σε ποιο χρονικό ορίζοντα να υπολογίζουμε. Και το Δεκέμβριο ε, ρώτησα και το Συμβούλιο. Και αυτό είναι θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τη χώρα μου και την κυβέρνησή μου. Εσείς με την ησυχία σας θα ήθελα και πάλι να σας πω ότι η συμπροματική ερώτηση αυτή δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη. Συμπροματική ερώτηση είπαμε, όχι καινούρια. Ε, αλλά εν πάση περιπτώσει απαντήστε, κύριε Ντοκούκτ. Ε, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω έκανε έκθεση για την παιδική εργασία. Η έκθεση αυτή είναι έτοιμη και συντομότατα θα διαβεβαστεί στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Εξ όσων γνωρίζω όμως, όλα αυτά θα συμβούν ακόμα ε, κατά την παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι αρμόδια κυρία Φεραίρο Βάλτνερ. 27 Ιανουαρίου λίγη η θητεία που είναι και τα γενέθλιά μου κατά τα άλλα. Thank you. Now I give the floor to Mr. Zalewski from the EPP. Ο κύριος Ζαλεύσκη από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων και ε, δίνει νέε αρμοδιότητες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ξένες επενδύσει. Πώς θα χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που προέρχονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας για να προασπίσετε τα οικονομικά και επενδυτικά συμφέροντα των ε, μεμονωμένων κρατών μελών σε περίπτωση που παραβιάζονται από τις δραστηριότητε των τρίτων χωρών. Δεν μιλάω μόνο για τους τελωνιακούς φραγμούς, αλλά και τους μη τελωνιακούς φραγμούς που στρέφονται εναντίον συγκεκριμένων ε, κρατών μελών. Το ίδιο αφορά τις επενδύσεις σε τρίτες χώρες από εταιρείε διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών μελών. Ε, για πολιτικούς λόγους χώρες όπως η Ρωσία, ας πούμε, μπορούν να έχουν συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένη στάση που παραβιάζει τα συμφέροντα. Ε, η επένδυση είναι οι επενδύσεις είναι καινούργια αρμοδιότητα τη εμπορική πολιτικής. Διευρύνονται οι αρμοδιότητές μας και αυτό είναι σημαντικό. Ε, θα πρέπει να δούμε την εμπορική εικόνα ε, μέσα στο ευρύτερό τη πλαίσιο και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε περισσότερα προβλήματα. Και θα πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή μια ευρεία συζήτηση βάσει της ανακοίνωση ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν ε, σημερινέ επενδυτικέ συμφωνίες για την προστασία των επενδύσεων. Υπάρχουν χιλιάδε τέτοιε συμφωνίες. Δεν πρόκειται να τις καταργήσουμε. Θα τις διατηρήσουμε, θα, διατηρήσουμε, θα εξασφαλίσουμε μια ασφάλεια δικαίου και θα προβούμε σε κάποιες πρωτοβουλίες και εμείς αλλά και κάποιες χώρες θα πρέπει να προβούν σε κάποιες πρωτοβουλίες για τις επενδύσεις, ε, θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τις επενδύσεις στις τρίτες χώρες. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σύντομα. Ε, συνδέεται και με την ενεργειακή ασφάλεια. Πρόεδρε, θα μπορούσα να... Έχω να πω περισσότερα, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω το χρόνο, δεν μου δίνετε το χρόνο. Κύριος Ζαλεύσκη συνεχίζει το δεύτερο ερώτημά μου. Ε, το δεύτερο ερώτημα συνδέεται με το πρώτο και αφορά την προστασία του ελευθέρου εμπορίου και τη χρήση του ελευθέρου εμπορίου για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών. Μιλήσατε για την Ουκρανία, μιλήσατε για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Ουκρανία. Πιστεύετε ότι αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία, θα πρέπει να είναι εντελώς αυτόνομη και δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εσωτερική κατάσταση της χώρας αυτής ή το αντίθετο. Αν δώσουμε κίνητρα στην Ουκρανία, αν της δώσουμε υποφελείς ε, λύσεις, δεν την ενθαρρύνουμε με αυτόν τον τρόπο για να συνεχίσει την ε, μεταρρυθμιστική της προσπάθεια, για να αναπτύξει και μια ελεύθερη αγορά και ένα κράτος δικαίου. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή με την Ουκρανία λέει ο Επίτροπο, είναι τμήμα ενό ευρύτερου πακέτου που προϋποθέτει και κάποια πολύ σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ε, είναι σημαντική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, γιατί είναι προτεραιότητα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη, σε αυτή τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου θα πρέπει να έχουμε διατάξεις, και είναι σημαντικό, γιατί τις εργασιακές σχέσεις, για το εργατικό δυναμικό. Διατάξεις επίσης για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Δηλαδή δεν πρόκειται για μια απλοϊκή προσέγγιση που να εστιάζει μόνο στο εμπόριο. Ε, έχει τα συνηθισμένα θέματα που έχουμε σε αυτές τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, όπως αυτά που περιλαμβάνει και η συμφωνία ας πούμε, με την ε, Κορέα. Αλλά βεβαίω η ενέργεια στην περίπτωση τη Ουκρανία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι σημαντική για την ε, ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τη Ευρώπη. Ο κύριο Κούτα από του Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα σημαντικό θέμα θα ήθελα να συζητήσουμε. Το αναφέρατε κι εσεί, ε, κύριε υποψήφιο επίτροπε, στην αρχική σα παρέμβαση, αλλά δεν επανήλθατε. Θα ήθελα να σα δώσω τώρα την ευκαιρία να πείτε λίγα λόγια παραπάνω. Μιλάω για το σεβασμό του περιβάλλοντος, για τα δικαιώματα των, του εργατικού δυναμικού και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Τι έχετε να πείτε για την αυτόματη συμπερίληψη αυτών των κριτηρίων στις ε, διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Συμφωνείτε. Αυτόματη συμπερίληψη, ε, αν ε, εννοείται ότι θα τα αντιμετωπίσουμε, προφανώς θα τα αντιμετωπίσουμε και φυσικά θα απεικονίζονται στις συμφωνίες. Από την άλλη όμως δεν πιστεύω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για αυτόματη συμπερίληψη με την έννοια δηλαδή ότι οι διατάξεις αυτές θα είναι ταυτόσιμες σε όλες τις συμφωνίες. Γιατί ο βαθμός ανάπτυξης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπορική μας πολιτική για να προωθήσουμε τις αξίες μας. Πρέπει να κάνουμε και μια προσπάθεια έτσι ισορροπίας, λεπτής ισορροπίας. Με το εμπόριο μπορούμε να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες αυτές, στους εμπορικούς μας εταίρους. Αυτό δεν γίνεται αυτόματα όμως, θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Σίγουρα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε κάποιες αναφορές στις συνθήκες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και ότι ο μη σεβασμός αυτών των ε, συνθήκων θα πρέπει να έχει κάποιες ε, επιπτώσεις. Επίσης θα πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον. Θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ανάλογα με, το, με τη χώρα και θα πρέπει να είναι όλα αυτά τμήμα των διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτές οι συμφωνίες παραμένουν εμπορικές και η ιδέα από πίσω είναι ότι προωθείται το εμπόριο. Αλλά με σεβασμό των στοιχείων που μόλις αναφέρατε. Άλλη ερώτηση, παραμένω στο ίδιο θέμα. Θα ήθελα να συνεχίσετε. Να υπενθυμίσω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε το 2009 ε, έχουν ε, ενεργοποιήσει έναν εμπορικό νόμο ε, που προτείνουν να ενταχθούν αυτά τα στοιχεία στις ε, δικές τους συμφωνίες. Η Κομισιόν τι θα κάνει ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει σε μια νέα εμπορική τροχιά στο σημερινό κόσμο. Απάντηση. Για αυτά τα θέματα η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την ίδια προσέγγιση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και αυτέ κινούνται προ την κατεύθυνση τη συμπεριλήψη όλων αυτών των κριτηρίων στι συμφωνίε. Αλλά όχι μόνο να τα συμπεριλάβουν, να συμπεριλάβουν αυτά τα κριτήρια, αλλά να τα συμπεριλάβουν με έναν τρόπο που να έχουν ουσιαστική επίπτωση. Ε, με αυτό διευκολύνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει το ίδιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εμπόριο σημαίνει και ανταγωνισμό. Ανταγωνισμό μεταξύ των εμπορικών εταίρων και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε να έχουν την ίδια προσέγγιση. Μην ξεχνάτε ότι μαζί είμαστε πάνω από το 50% της παγκόσμιας οικονομίας. Αν λοιπόν, αν θέλουμε να θέσουμε ε, πρότυπα, πρέπει να τα θέσουμε από κοινού. Και τώρα, ο κύριος Φάβα. από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σάλμπα, ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω στην Κορέα. Είπατε κύριε υποψήφιοι επίτροπε. Ορισμένα μέτρα όπως το duty pack που ε, ανησυχούν πολύ την αυτοκινητοβιομηχανία ή την κλωστοϊφαντουργία δεν είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με το μέγεθος της χώρας αλλά με την ανάπτυξή της και το βιωτικό επίπεδο. Προσοχή, προσοχή, γιατί αυτό συνιστά σημαντικό προηγούμενο και το τονίζω, σημαντικό προηγούμενο σε μελλοντικέ συμφωνίες με άλλες χώρες που κρατούν άλλες συνθήκες και έχουν και διαφορετικό μέγεθος. Πολύ σημαντικό αυτό και θέλω να μάθω και την άποψή σας. Στη συνέχεια, στρατηγική ε, σχέση με τη Λατινική Αμερική. Στην εμπορική πολιτική, στη συμφωνία την εμπορική με την Κεντρική Αμερική που περίπου έχει λήξει ε, αν λυθεί το, αφού λύθηκε το θέμα μάλλον της μπανάνας των ΠΟΕ και ε, θεωρήθηκαν ε, ανώθευτες οι εκλογές του Νοεμβρίου στην Ονδούρα θα προωθηθεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την παρατήρησή σας για το duty drawback για τη μείωση των δασμών. Σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να δοθεί σημασία σε αυτό το θέμα. Πάντως αυτό το θέμα δεν εμφανίζεται δεν εμφανίστηκε έθνης, ας πούμε, στη Συμφωνία Ελευθερίου με την Κορέα. υπάρχει και στην σημερινή συμφωνία με την Κολομβία. Δεν είναι μία καινοτομία, λοιπόν. Θα πρέπει να δώσουμε σημασία. Για την Λατινική Αμερική υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα και είναι η Ονδούρα. Είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε απέναντι στην Κεντρική Αμερική παρουσία και της Ονδούρας θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή υπάρξει κυβέρνηση. Αλλά είναι μια πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί. Και εκεί θα πείτε κι εσείς ε, την άποψή σας. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε. Το θέτω και σε εσά. Θα διαπραγματευτούμε με αυτούς ή όχι. Δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Επίση, αναφερθήκατε στην Κολομβία και είπατε ότι υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα και ρήτρα. Όπω γνωρίζετε όμω, και υπάρχει περίπτωση να μην είναι τόσο ισορροπημένη η ε, συμφωνία. Ε, αν πρέπει να περιμένουμε πέντε χρόνια για να κινητοποιηθεί αυτή η ρήτρα, μπορεί να είναι πολύ αργά για την Κορέα. Ρωτάτε για την Κολομβία. Για την Κορέα, ναι, ναι. Υπάρχει αυτό το μέτρο για την επιστροφή του δασμού και τίθεται σε ισχύ πέντε χρόνια μετά. Και εγώ έθεσα το ερώτημα γιατί. Η απάντηση είναι ότι αυτή είναι η στιγμή που δεν υπάρχουν πια δασμοί. Αρχίζει να ισχύει μόνο όταν δεν υπάρχουν πια δασμοί. Γιατί αν υπήρχαν δασμοί θα υπήρχε αντίφαση. Ελπίζω να απαντάω στο ερώτημά σας. Κύριε Ντεσαρνές, από το Άλντε, τους φιλελεύθερους. Είπατε κατ' επανάληψη ότι για σας το διεθνές εμπόριο δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά θα πρέπει να είναι εργαλείο ε, στα χέρια της πολιτικής που θέλει να πετύχει κάποιους στόχους. Καλό αυτό. Α, αλλά θα πρέπει εν διάφορη περιπτώσει να προωθήσετε κάποιες μεταρρυθμίσεις, κάποιες αλλαγές. Είσαστε έτοιμοι να, ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσετε κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποίησεις των ΠΟΕ, να υπάρξουν κάποιοι κοινωνικοί, υγειονομικοί κανόνες, κανόνες καλής διακυβέρνησης. Είσαστε έτοιμοι να φτάσετε μέχρι εκεί. Έχετε αυτό πνεύμα μεταρρύθμισης ή όχι. Επίσης είπατε ότι αυτό το φόρο για τον άνθρακα α, δεν μπορούμε με, με μιας έτσι να τον καταργήσουμε. Θα ήθελα η Μελλοντική Επίτροπη να μας ε, πει θα ξεκινήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα μία μελέτη αντικτύπου και συνεχεία θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αυτό που είπα είναι το εξή. Είπα ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στον ΠΟΕ και να συζητήσουμε για αυτές αυτή στιγμή ολοκληρωθεί ο γύρος της Δόχα. Δεν έχει νόημα να γίνει τώρα. Τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το γύρο και εν συνεχεία να δούμε τι θα κάνουμε με τα ερωτήματα που θέσατε για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάνω απ' όλα τα κλιματικά ζητήματα, τα κλιματικά προβλήματα που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές. Σε ό,τι αφορά το φόρο για τον άνθρακα, για το διοξίδιο του άνθρακα δηλαδή. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Και εσείς το ζήσατε στη χώρα σας. Γιατί υπήρχε ένα φόρο ε, για το διοξείδιο του άνθρακα και το συνταγματικό σας δικαστήριο τον ακύρωσε γιατί δεν σεβόταν την ε, αρχή της νομιμότητας. Το ίδιο πρόβλημα θα τεθεί και στο μέλλον. Φαντάζομαι λοιπόν θα παρουσιαστεί μια αναθεώρηση αυτού του, νομος, του νόμου. Θα πρέπει καταρχάς λοιπόν να υπάρχει ε, σεβασμός της αρχής της νομιμότητας. Είμαι πεπισμένος όμως ότι αν γίνει αυτό θα υπάρξει μια πλειοδοσία και θα φτάσουμε σε εμπορικό πόλεμο. Δεν νομίζω ότι το οικονομικό μας σύστημα εξυπηρετείται με ένα τέτοιο φόρο. Πριν κάνουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ. Μιλήσατε για μια μελέτη αντικτύπου. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι ξεκίνησε μια τέτοια μελέτη. Πρέπει να το τσεκάρω με τις υπηρεσίες μου. Α, το θέμα δεν είναι να, δούμε, να κάνουμε μια μελέτη αντικτύπου όμως, αλλά θα πρέπει να δούμε και κατά πόσο πρέπει να κάνουμε μια μελέτη σκοπιμότητας. Νομίζω ότι πρέπει να αξιολογήσουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για αυτό το θέμα μπορούμε να κάνουμε μια, μια μελέτη. Και για το θέμα της ανάπτυξης. Είσαστε αυτή τη στιγμή ε, επίτροπος ανάπτυξης. Πιστεύω ότι το ε, αποτέλεσμα της εμπορικής πολιτικής και της αναπτυξιακής πολιτικής για τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι θετικό. Δεν νομίζω ότι το άνοιγμα, πάση θυσία των αγορών εξυπηρετεί το, τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε τρομερές ανισότητες, αύξηση στις, στις ιδίω ιδίως στις φτωχέ χώρε όπω στην Αφρική, που δεν, μπορεί άνθρωπο, δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν από τη γη του. Θα πρέπει να δούμε ξα, ξανά τι διακυβεύεται ε, για τι αναπτυσσόμενε χώρε με την εμπορική πολιτική. Πρέπει να το, την ξαναδούμε άρδιν. Ίσως θα πρέπει να την ανα, μεταρρυθμίσουμε εκ θεμελίων τα επόμενα χρόνια. Ένα λεπτό αυστηρά για αυτήν την απάντηση. Και, στο, και εγώ στο παρελθόν και στους τελευταίους αυτούς μήνες σκέφτηκα πολύ σοβαρά τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στις ομενες χώρες. Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Από την άλλη, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ο, ο και ο ένοχος ο γύρος της Ντόχα και ο ΠΟΕ. Όταν εξετάζουμε τις ε, λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες δεν μειώνουν και δεν χρειάζεται να, μειώσουν τους εδασμού του στο γύρο τη Ντόχα. Κι όμως αυτές οι χώρες τι ευρωπαϊκέ αγορέ, έχουν ελεύθερη πρόσβαση. Ε, στα πλαίσια του μηχανισμού όλα πλην όπλων. Είμαστε οι μόνοι που του δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θέλουμε να γίνει και ευθύ ε, στο γύρο τη Ντόχα. Δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι το οποίο φύγει τα συμφέροντα των χωρών αυτών. Μην ξεχνάμε όμως ότι η ανάπτυξη είναι ένα περίπλοκο θέμα και το συνειδητοποιώ όσο περνάει ο καιρός. Και τώρα δίδω το λόγο στον κύριο Φιέλνερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς χαίρομαι που ακούω ότι θέλετε να σεβαστείτε και να ε, τηρείτε τις υποσχέσεις στο εμπόριο, στο παγκόσμιο εμπόριο. Πέρα από τους κινδύνους του προστατευτισμού έχουμε και κινδύνους για το περιβάλλον. Μπορεί το εμπόριο να χρησιμοποιηθεί όμως και σαν ευκαιρία, όχι μόνο σαν απειλή να θεωρείται για το περιβάλλον. Μπορούμε να βρούμε κάποιες μεθόδους για να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα του περιβάλλοντος με περισσότερο εμπόδιο. Εμπόριο, συγγνώμη. Στην Κοπενχάγη πολλοί θέλαν να θέσουν νέα εμπόδια στο εμπόριο αντί να το απελευθερώσουν. Και αυτό ενέχει το κίνδυνο της αποτελμάτωσης, της καταπολέμησης, της ένδυας. Πώς μπορούμε λοιπόν με περισσότερο εμπόριο να λύσουμε τα περιβαλλοντικά θέματα. Φοβάμαι ότι τώρα θα πρέπει να γίνω πιο αυστηρός γιατί έχουμε καθυστέρηση 10 λεπτών ήδη. Παρακαλώ για να απαντήσετε ένα λεπτό κύριε Ντεχάχτ. Ευχαριστώ. Μία από τις προσεγγίσεις που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε είναι να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε για πραγματικό ελεύθερο εμπόριο, για περιβαλλοντικά αγαθά, χωρίς δασμούς. Κατάργηση των δασμών. Κάναμε πρόταση Προφανώς του παρόντος αυτό είναι αδύνατο σε επίπεδο ΠΟΕ, αλλά προσπαθήσαμε να ε, αναστήσουμε κάποια συμμαχία αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες ε, για να μπούμε σε ένα τέτοιο σχήμα. Βέβαια υπάρχουν και δυσκολίες άλλου είδους. Για παράδειγμα, η Βραζιλία θέλει να βάλει στη λίστα τη βιοεθανόλη ως περιβαλλοντικό προϊόν. Αλλά αυτό χρειάζεται μεγάλη συζήτηση, γιατί υπάρχουν διαφορετικά είδη βιοεθανόλης, δεν είναι όλα η φόρα προϊόντα και η κατάργηση των δασμών για περιβαλλοντικά προϊόντα έχει να κάνει με παραγωγή και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και τεχνικές και μεθόδους. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να το μελετήσουμε πολύ και υπάρχει και ο ΠΟΕ που μας ε, περιορίζει κάπως. Συμπροματική ερώτηση, ο κύριος Φιέλνερ. Ευχαριστώ. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια αντίστοιχη ε, συμφωνία όπως έχουμε για την πληροφορική ας πούμε και για το περιβάλλον. Με ικανοποιούν αυτό που μας λέτε. Τι γίνεται όμως με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία, γιατί έχουμε νέους φραγμούς πλέον μη δασμολογικούς και θα ήθελα να μάθω την άποψή σας. Εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευρωπαϊκή εμπειρία για να καταπολεμήσουμε αυτούς τους φραγμούς. Στο εσωτερικό της Ευρώπης το λύσαμε και έτσι δεν έχουμε ανεπιθύμητα εμπόδια στο εμπόριό μας. Δεν θα μπορούσαμε αυτό να το μεταφέρουμε και ε, στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που έχουμε με άλλες χώρες και σε μερές επίπεδο. Έτσι ώστε ακριβώς οι κανόνες για το περιβάλλον να μην σημάνουν νέα άσκοπα και άχρηστα εμπόδια στο εμπόριο. Όταν προσπαθεί κάποιο να φτιάξει μια αγορά, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι καταργεί του δασμού. Αυτό κάναμε και στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή σε εξαφανιστούν λοιπόν οι δασμοί, έχουν την τάση να αναδύονται και να εμφανίζονται περισσότερο και με πιο μεγάλη περιπλοκότητα ε, άλλοι φραγμοί, μη δασμολογικοί. Το είδαμε και στην Ευρώπη και χρειάστηκε μια δεκαετία για να τους καταργήσουμε. Και μάλλον θα χρειαστεί και περισσότερος χρόνος διεθνώς. στον ΠΟΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε πάντως υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν εγκρίνεται μια νομοθεσία, δεν θα πρέπει να έχει παρενέργειες. Γιατί καμιά φορά δεν είναι παρενέργειες, είναι επίτηδες και μένει για να δημιουργούνται τέτοια εμπόδια καινούργια. Και πολλές φορές βλέπουμε από την περιβαλλοντική νομοθεσία ότι τελικά είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευτική. Αλλά αυτό δεν είναι καινούριο. Παρατηρείται σε κάθε είδους νομοθεσία και γιατί να μην συμβεί και με την οικολογική νομοθεσία. Άλλωστε. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λάγκε από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντεχόχτ, συμφωνούμε πιστεύω ότι η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να ε, θέτει ένα αμφιβόλο τα κεκτημένα στην Ευρώπη και το κοινωνικό πρότυπό μας και το βαθμό ελευθερίας μας. Παράδειγμα, το πακέτο των τηλεπικοινωνιών. Πριν από μερικούς μήνες αποφασίσαμε την προστασία των χρηστών του διαδικτύου για να τους ε, προστατεύουμε από περιορισμούς και από αποκλεισμούς και έγινε και εντονότατη αντιπαράθεση. Τώρα ακούω για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε ότι τίθεται ένα αμφιβόλο αυτό το κοινοτικό μας και εκτιμένο. Είναι οι διαπραγματεύσεις άκτα. Μπορείτε εσείς να μας εγγυηθείτε ότι δεν θα αναβαγίσει το πακέτο των τηλεπικοινωνιών, θα προστατεύεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο και θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις που έχουμε τώρα και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Κοιτάξτε για τη διαφάνεια έχω ήδη απαντήσει σε μία από τις πρώτες ερωτήσεις. Είναι προφανές ότι θα σεβαστώ τη διαφάνεια. Θα επιμείνω στη δέσμη των τηλεπικοινωνιών στο ΆΚΤΑ. Το ΆΚΤΑ δεν σκοπεύει να είναι κλειδί που θα κλείσει την πόρτα στο Ιντερνετ, όχι. Αλλά οι απομιμήσεις να καταπολεμούνται. Και όχι μόνο οι οργανωμένες απομιμήσεις από το οργανωμένο έγκλημα. Όχι το να φέρνει κάποιος ένα αγαθό απομίμησης στην Ένωση. Αυτό δεν μας. Συμπληρωματική. Ευχαριστώ. Και το δεύτερο είναι η κοινωνική μας συνοχή και συνύπαρξη. Και μιλάμε για εμπορικές σχέσεις με χώρες όπου επικρατούν άλλοι κανόνες με ντάμπινγκ στους μισθούς ή απαγορεύονται οι απεργίες όπως η Νότια Κορέα. τότε έχουμε μειονεκτήματα ε, ανταγωνισμού και πίεση που ασκείται στα κοινωνικά μας ε, συστήματα. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα ήδη στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τι συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να λάβετε για να διατηρηθούν οι προδιαγραφές και εργασίες και να προστατεύετε το κοινωνικό μας σύστημα. I'm really Λυπούμε που έχω μόνο ένα λεπτό αλλά θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερο εμπόριο για τη διατήρηση του κοινωνικού μας συστήματος προστασίας. Γιατί απαιτεί ανάπτυξη και είναι προφανές ότι η ανάπτυξη δεν θα, γίνει, δεν επιτευχθεί αυτόματα, ιδίως μετά την κρίση που ζούμε. Χρειαζόμαστε το εμπόριο. Τι να κάνουμε, έχουμε τα εργαλεία για την πρόθεση του εμπορίου, για την άμυνα του εμπορίου, θα τα χρησιμοποιήσουμε. δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τα χρησιμοποιήσουμε. Στη συμφωνία, η εμπορική συμφωνία με την Κορέα υπάρχουν ρήτρε για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σαφείς ρητέ παραπομπές στις συνθήκες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, παραδείγματος χάρη. Και αυτό θα ισχύσει όχι μόνο για την Κορέα αλλά και για την Κίνα. Η συμφωνία που πραγματευόμαστε με την Κίνα για την οποία δεν είμαι ο κύριος αρμόδιος, περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και θα τα προσέξουμε να γίνουν σεβαστά. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Παπαστάμκος από το ΕΛΚ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τις πιο ανοιχτές αγορές, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για πολλούς από τους εταίρους της που διατηρούν υψηλούς δασμούς παραδείγματος χάρη και οι εισαγωγές προς την Ένωση σημειώνονται πολλές, στις εισαγωγές σημειώνονται πολλές φορές φαινόμενα κοινωνικού και περιβαλλοντολογικού dumping. Αυτό δεν αποτελεί μόνο ε, ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, αλλά μπορεί να αποτελέσει και κίνδυνο για τους καταναλωτές. Τι θεωρείτε λοιπόν τις απαραίτητες ε, παραμέτρους μέτρα της Ένωσης για να μπορέσει να εξισορροπηθεί το πρόβλημα πολύπλοκο το ερώτημα για το γύρο της Ντόχας πρέπει να δούμε ποια είναι η φύση του. Είναι αναπτυξιακός. Πρέπει λοιπόν το αποτέλεσμα να εξυπηρετεί ακριβώς το στόχο αυτό, δηλαδή τις αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες να καταστά δυνατόν να γίνουν τμήμα της διεθνούς οικονομικής ζωής. Αυτό είναι ουσιώδες και η Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτήν ακριβώς τη θέση παίρνει αποφασιστικά στις διαπραγματεύσεις. Εξάλλου δεν είναι μόνο πρόβλημα του, αλλά και νότου νότου. Και υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών, κατηγοριών αναπτυσσομένων χωρών. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις βοηθήσουμε πάντως. Επίσης θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται πάντοτε εξισορρόπηση από τη μία μεταξύ της επιβολής κριτηρίων που θα ήταν πιο φυσικά μέτρα μέσα στην Ένωση και από την άλλη της ευκαιρίας που πρέπει να δοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες για να είναι οικονομικά ενεργές. Και γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες μέτρων. Πρέπει να επιτεθεί μια συμφωνία και εγώ νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε αλλά να μην αγνοούμε επίσης τις βαθμούς διαφοροποίησης. Δεύτερη ερώτηση. Η προηγούμενη Επίτροπος είχε μιλήσει για σφαιρική πρόσβαση στις αγορές και τη στρατηγική που την αφορά. Ποιο είναι το σχέδιό σας για να βελτιωθεί το περιβάλλον, το κλίμα εφαρμογής ελεύθερης αλλά και δίκαια, ε, ελεύθερο και δίκαιο διεθνούς εμπορίου. Παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο. Για την πρόσβαση στις αγορές. Την κάνουμε για να αμυντικά αλλά πρέπει να την εφαρμόσουμε επιθετικά δηλαδή. Σημειώστηκαν ορισμένες επιτυχίες πρόσφατα ως την πρόσβαση της αγορές για την Αίγυπτο και τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό είναι αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής μας, η καταπολέμηση δηλαδή μέσα στα νομισμένα πλαίσια των προβλημάτων που αφορούν τους μη τελωνιακούς δασμούς ιδίως, δε φραγμούς ιδίως. Τώρα η κυρία Ντεκέιζερ, σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιούμε και την ειλικρίνειά της. Είναι πια παρημιώδης η ειλικρίνειά σας και με τα τελευταία συμβάντα στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό φάνηκε ότι οι αρχές της καλής διακυβέρνησης, της κοινωνικής δικαιοσύνης κλπ είναι κάτι το αναπόφευκτο και σας υποστηρίζουμε στις ιδέες αυτές. Αλλά θυμάμαι το εξής ότι πρέπει όλα αυτά που είναι σωστά να εφαρμοστούν και όπως πρέπει. Ναι, το είπατε και εσείς το είπατε, δεν λέω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μεν κάποια, κάποιος έλεγχος των ζημιών που μπορεί να προκληθούν από υπερβολικά ελεύθερο εμπόριο, αλλά είναι αυτό το τμήμα της στρατηγικής σας. Ας μην κάνουμε συζήτηση μεταξύ Βέλγων, κυρία Ντεκέιζερ. Αυτά που είπα στις 16 Δεκεμβρίου εδώ είχαν γίνει δεκτά ομόφωνα και από την πολιτική σας ομάδα. Μα ναι, για κομπλιμέντο σας τα είπα. Α, ναι, α, δεν το είχα καταλάβει. Α, καλά τότε, καλά. Εγώ προσπαθώ απλώς να είμαι συνεπής, Δεύτερη ερώτηση, Βερόνικα. Ναι, φυσικά, φυσικά συνεπής. Νομίζω ότι, για, επιμένω, σας το είπα για κομπλιμέντο, αλλά εννοώ ότι εσείς εξηγηθήκατε ως προς το τι θα κάνετε για την Κολομβία, αλλά οι αρχές της καλής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπά πρέπει να εφαρμοστούν και εκεί και απλώς θα θέλαμε και εκεί να φανείτε συνεπείς. Αυτό είναι και αποτελεσματικό. Μα δεν ήταν ερώτηση, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω σας τα εξήγησα. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Κολομβία, τίθεται σε πολλές συμφωνίες που πρέπει να συνάψουμε. Η κατάσταση βέβαια είναι πάντα διαφορετική, αλλά γι' αυτό είναι ακριβώς είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνέπεια. Ευχαριστώ. Και τώρα έχω τη χαρά να δώσω το λόγο στην κυρία Μουσκαρδίνη, συνάδελφο αντιπρόεδρο από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πίσω σας είμαι κύριε Μπεχούχτα. Ε, είσαστε και προετοιμασμένος και επαΐων. Αλλά η απάντηση που δώσατε στην κυρία Σαΐφη και σε άλλους συναδέλφους για το θέμα του ντάμπικ ε, εστράφει γύρω από την Τόχα. Ξέρουμε ότι εδώ και χρόνια μας λένε ότι θα ολοκληρωθεί και θα τελεσφορήσει, αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης και στις γραπτές σας απαντήσεις ε, μιλήσατε για τον ΠΟΕ. Ε, από αυτά που μας είπατε εδώ προφορικά και από τα γραπτά σας σχόλια, ε, προκύπτει ότι πιστεύετε στη συνεργασία μεταξύ ημών και, και εσάς κύριε Επίτροπε. Ε, για το θέμα της ονομασίας των εμπορικών σημάτων. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί ένα τμήμα του Συμβουλίου δεν συμφωνεί. Αλλά όμως δεν μας είπατε πώς θα προχωρήσετε εσείς. Δεν δεσμευτήκατε καθόλου. Μιλάω για το πρόγραμμα του Οκτωβρίου της Επιτρόπου Άστον. Η Ιταλία είναι μία από τη χώρα, λέει ο Επίτροπος, όπου το θέμα αυτό συζητείται. Και είναι κατανοητό αυτό. Και εσείς όμως πρέπει να καταλάβετε ότι μπορούμε να έχουμε μια τέτοια νομοθεσία μόνο εφόσον συμφωνήσει το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο, γιατί αυτό είναι το τμήμα της συναπόφασης. Η κάθε Άστον έκανε κάποιες προτάσεις και προσπαθεί να ξεφορτωθεί τα, προβλήματα, τα σημεία που δημιουργούν πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό να έχουμε τέτοιο κανονισμό. Θα προσπαθήσω για κάτι τέτοιο. Αλλά το Συμβούλιο είναι μπροστά μας. Ε, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει συμφωνία ε, γιατί υπάρχει διχασμό στο Συμβούλιο. Ε, αρκεί μια πλειοψηφία. Χρειάζεται μια πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Θα προσπαθήσω να δημιουργηθεί αυτή η πλειοψηφία καλό θα ήταν να με ρωτήσετε το ίδιο πράγμα μετά από λίγους μήνες, όταν θα έχω και μεγαλύτερη εμπειρία με το συγκεκριμένο θέμα για τα εμπορικά σήματα. Πολύ ωραία. Καταγράφω τη καλή σας θέληση. Το να περιμένουμε μήνε, κάποιους μήνες είναι υπερβολικό. Θα θέλαμε να γίνει προσπάθεια σύντομα, ούτως ώστε και εμείς το Κοινοβούλιο μαζί με την Κομισιόν να δούμε τι θα κάνουμε απέναντι στο Συμβούλιο. Γιατί αλλιώς η συναπόφαση ε, είναι μόνο επί χάρτου. και η συνεργασία ε, Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν δίνει αποτελέσματα. Για την ονομασία προέλευσης και για την πρόταση κανονισμού θέλετε να κάνετε μια προσπάθεια για να εναρμονίσετε τα λεωνιακά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών μια και ε, υπάρχουν προβλήματα με απομιμήσεις προϊόντων που εισάγονται. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να αντιμετωπίσουμε τα ψευδεπίγραφα προϊόντα με ένα κοινό πρόγραμμα. Ε, επίσης, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, το σχάρι, τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Ε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα θέματα. Απάντηση για τον κανονισμό. 1383 για τα τελωνιακά θέματα. Θα αναθεωρήσουμε τον κανονισμό αυτού του 2003. Γιατί στην Ολλανδική περίπτωση ε, το θέμα αφορούσε τα γενώσιμα φάρμακα. Και αυτός ο κανονισμός εφαρμόστηκε. Όχι με φυσικό τρόπο για να το πω έτσι. Ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε, να χτενίσουμε αν θέλετε αυτόν τον κανονισμό. Για να δούμε πώς μπορούν να εξάγονται χωρίς εμπόδια τα γενώσιμα φάρμακα. για τον κανονισμό. Ο κανονισμός ε, αποφασίζεται με συναπόφαση. Δεν μπορείτε να πείτε ότι αυτό είναι απλά λόγια, λόγια και ένα περιεχομένο. Είναι μια διαδικασία με καθυστερήσεις, με πρωτοβουλίες ενδεχομένω από τα συμμετέχοντα όργανα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, με διαδικασίες ε, συνδιαλλαγής και με αποτελέσματα. Ε, και εγώ θα προσπαθήσω να διευκολύνω τη διαδικασία, αλλά δεν συμμετέχω στην πραγματικότητα στη διαδικασία ε, συνδιαλλαγή. Είναι θέμα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου να συμφωνήσουν τελικά. Κυρία Λούκα, από του Πράσινου. Ε, εκ μέρου ενό συναδέλφου που είναι απόν. Ε, ο κύριος Λάγκερ μίλησε για τις συμφωνίες ε, εμπορίου κατά καταπολέμησης των ψευδεπίραχων προϊόντων. Δεν θα πρέπει να εστιάσουμε πάλι στη διαφάνεια. Ε, το Κοινοβούλιο το έχετε κρατήσει στο περιθώριο από αυτές τις συζητήσεις. Δεν είδαμε ποτέ τα προσχέδια των διαφόρων κεφαλών. Η Γενική Διαθέση ε, Εμπορίου λέει ότι υπάρχει θέμα εμπιστευτικότητα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το ζήτησαν, είπα, γιατί δουλεύουν με τους κανόνες της γρήγορης διαδικασίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφορετικέ διαδικασίε, διαφορετικό νομικό πλαίσιο. Ε, με τη διαδικασία τη Λισαβόνα, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, δώσει τη γνώμη του. θα πρέπει να εμπλακούμε. Πώ θα ενημερώσετε το Κοινοβούλιο, όπω ενημερώνεται το Συμβούλιο για τι διαπραγματεύσει, ούτω ώστε να υπάρχει δυνατότητα να εκφράσουμε τι απόψει μα και να ληφθούν, να ληφθούν από εσά υπόψη οι συστάσει μα. Και επίση σε ποια φάση mm. της ε, διαπραγμάτευσης θα διαβιβάσετε τα στοιχεία στο Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνω τις ε, ε, ανάγκες περιεμπιστευτικότητας, αλλά πρέπει να καταλάβετε κι εσείς τα νέα δεδομένα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αν υπάρχει μια διαδικασία εμπιστευτικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων μερών, θα πρέπει να τη σεβαστώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε μια πλήρη συζήτηση για τις κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είσαστε, να είσαστε ήσυχοι ότι θα λάβω υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά όταν μπαίνουμε ε, σε μια διαπραγμάτευση η οποία είναι εξελίξη, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες. Εγώ θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω ε, θα προσπαθήσω να δώσω την ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις σας και να τις λάβουμε υπόψη βέβαια. Η επόμενη ερώτηση. Τότε δεν ξέρω αν κάνατε καλά που δεχθήκατε αυτούς τους όρους ε, ε του απορρίτου της εμπιστευτικότητας. Ξέρω ότι δεν ήσασταν εσείς, αλλά το κοινοβούλιο θα πρέπει να παίζει πλήρη ρόλο σε μια τέτοια συζήτηση, έτσι δεν είναι. Και υπάρχουν νομικά κολλήματα, θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε πλήρη πληροφόρηση. Ερώτηση. Θα έπρεπε να είχε γίνει καν αυτή η συμφωνία για την εμπιστευτικότητα. Και τι γίνεται με τη Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορίου με τον Καναδά που επίκειται. Έχει και αυτή τέτοια στοιχεία απορρίτου και εμπιστευτικότητα. Δεν ξέρω. Ε, μπορεί να τα βρούμε διαφορετικά με τον Καναδά και να μην είναι απόρριτη η συμφωνία. Θα γνωρίζετε ίσως ότι έχετε νέες αρμοδιότητες τώρα ε, για το εμπόριο και είναι πραγματικά ολοκένουργες. Ναι. Ε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχετε δικαίωμα απόφαση πλέον ε, και σύμφωνης γνώμης για τις συνθήκες. Είναι πολύ φρέσκες αυτές οι αρμοδιότητες. Οπότε αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητας παραχωρήθηκε με βάση το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε που ήταν τελείως διαφορετικό ή στο εξή θα πρέπει κάθε φορά να εξετάζουμε και να κρίνουμε αν χρειάζεται τέτοια εμπιστευτικότητα. Και φαντάζομαι θα κάνετε και εσείς τέτοιες ερωτήσεις αντίστοιχες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι καμιά φορά για να γίνουν διαπραγματεύσεις καν θα πρέπει να εξασφαλίζονται ορισμένες συνθήκες απορρίτου και εμπιστευτικότητα. Είναι μια πάρα πολύ λεπτή ισορροπία και άσκηση που θα πρέπει από κοινού να ε, κάνουμε σε σχέση με τον Καναδά τώρα όμως είναι νέο το καθαστώς, επαναλαμβάνω και θα εξασφαλίσω πλήρη σας συμμετοχή ωστόσο Μιλάμε πάντα για διμερή συμφωνία, έτσι, και θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Είναι άλλο το πλαίσιο από την πολυμερή συμφωνία. Now Και τώρα και πάλι ο κύριος Σάχραντι, εξ ονόματος της ομάδας των συντηρητικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τρίτη φορά παίρνω το λόγο, αλλά και τελευταία. Φτάνει πια τρεις φορές. Σε ό,τι αφορά αυτή την πίεση που ασκούμε για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικές σχέσεις, καλό είναι, αλλά έχουμε και το αντίθετο φαινόμενο. Παράδειγμα, η Σρι Λάνκα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι. πρότεινε αναστολή του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ακριβώς για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Και είδαμε ότι αυτό ε, βοήθησε και βελτιώθηκε δραματικά η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι χάρη στη δική μας πίεση. Λοιπόν, ακριβώς επειδή μπορεί να έχει και θετικό αποτέλεσμα όπως είδαμε στη Σιλάνκα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Κοιτάξτε, σας πω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια βαθύτατη ανάλυση των ε, γεγονότων. Καταλήξαμε ότι τρεις παρακαλώ συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας δεν γίνονται σεβαστές. Προτείναμε στο Συμβούλιο να λάβει αντίστοιχα μέτρα για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ, SPS+. Τώρα είναι επιτάπητο στο Συμβούλιο, έχουν ένα εξάμεινο για να το εξετάσουν και ε, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού θα συνεχίσουμε εμείς τις ε, επαφές και τις συνομιλίες με τη Σρι Λάγκα για αλλαγές που αναμένουμε σε σχέση με τις συμβάσεις ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Και ελπίζω να εκμεταλλευτούμε αυτό το εξάμεινο που έχουμε μπροστά μας για να βρούμε κάποιες λύσεις. Χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω μέτρα για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Πάντως, επί το παρόντες, έχουμε σοβαρούς λόγους να λάβουμε τα μέτρα αυτά και να πρόκειται στη Σρι Λάνκα να βελτιώσει την κατάσταση μέσα στο εξάμεινο που έχει στη διάθεσή της. Ευχαριστώ. Ακούσαμε και προηγουμένως να λέτε και σωστά λέτε, λέει ο κύριος Σάχραντιλ, ότι είναι σημαντικό να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπάρχει χρηστή διακυβέρνηση. Άλλο παράδειγμα, το Κονγκό χρόνια πόλεμο έχει. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες στην Αφρική, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναλλάστε με τις χώρες αυτές. Δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία που να μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε για να τους βοηθήσουμε. Να τους βοηθήσουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση του κράτους, να είναι καλύτερη διοίκηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχετε τίποτα τέτοιο υπόψη σας. Uh, αυτό το καιρό διαπραγματευόμαστε τις συμφωνίες οικονομικής εμπορικής σχέσης και προηγουμένως αναφέρθηκα στην ακρόαση σε αυτό. Θα πρέπει να είναι πάντα στο επίκεντρο το στοιχείο της ανάπτυξης για τις χώρες αυτές. αλλά και το εμπόριο έχει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Και μπορούμε να κάνουμε πολλές προσπάθειες για βοήθεια με σκοπό το εμπόριο. Aid for trade. Οι σχέσεις Αφρικής-Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν να κάνουν με τους δασμούς, γιατί δεν υπάρχουν δασμοί σε αυτές τις συμφωνίες ε, ε, είπα τα πάντα πλην όπλων, everything but arms. Ε, είναι θέματα επιμελητίας, είναι θέματα νομικού πλαισίου, αλλά όχι τελωνιακά. Και αυτό το συζητάμε πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπόριου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε καλύτερα στο μέλλον. Και περισσότερο. Ευχαριστώ. Και τώρα είναι η ώρα του κυρίου Ράμστορφ, εξ ονόματος της ε, Νοτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Εσείς και οι συνάδελφοί σας είστε καπετάνιοι ε, στη θύελα, στη φορτούνα και φορτούνα φουρτούνα σημαίνει οικονομική κρίση και η ανεργία ε, θα πλήξει πάνω από 57 εκατομμύρια ανθρώπους. Τεράστιο πρόβλημα στην Ένωση. Και ο καλύτερος τρόπος κατά πολέμησης της ανεργίας είναι η καινοτομία. 75% της ανάπτυξης του ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες χώρες συνδέεται με την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία. Ερώτηση λοιπόν, εσείς τι μπορείτε να κάνετε ως επίτροπος για να εφαρμόζετε καλύτερα, να μεταφέρετε καλύτερα η καινοτομία στην πράξη. Ε, μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι και να προσπαθήσει τουλάχιστον. Και είναι από τις βασικές αδυναμίες και λήψεις στην Ευρώπη αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται στην επανάσταση της μικροηλεκτρονικής. Οι σημαντικότερες εφευρές είναι μεν ευρωπαϊκές, αλλά οι βιομηχανικές τους εφαρμογές και η παραγωγή τους είναι σε μεγάλο βαθμό εκτός της Ευρώπης. Και θα πρέπει να φροντίσουμε, για παράδειγμα, για την πράσινη οικονομία να μην συμβεί το ίδιο. Δηλαδή, εμεί κάνουμε τις εφευρέσεις, την τεχνολογία και μας διαφεύγει η βιομηχανική παραγωγή, η εμπορική παραγωγή. Πώς θα γίνει αυτό, τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικέ ιδέες έχω, αλλά ρωτήστε καλύτερα άλλους συναδέλφου. Uh, Συμπροματική ερώτηση δεν ισχύει αυτό 100% που λέτε, διότι τα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά και το διεθνές εμπόριο είναι δική σας αρμοδιότητα. Και γι' αυτό σας ρωτώ. Και ψάχνω να βρω νέες μορφές παραγωγής, νέους τρόπους παραγωγής. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που είμαστε ε, ηγέτες στην ανοτεχνολογία, στην ανοεπιστήμη, στην οικολογική τεχνολογία και αυτά τα προϊόντα μπορούν να κυκλοφορήσουν στη διεθνή αγορά και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. τότε μιλάτε για το γενικό πλαίσιο του εμπορίου εσείς τώρα. Φυσικά έχουν, έχουν μεγάλη σημασία διαπραγματεύσεις για αυτά τα προϊόντα και για τα νάμα, τα μη γεωργικά και για τις υπηρεσίες. Είπα ήδη Είμαστε υπέρ της κατάργησης των δασμών για τα περιβαλλοντικά αγαθά. Και θα πρέπει να βρούμε μια συμφωνία. Το θέμα είναι πώς θα πουλήσουμε αυτά τα προϊόντα, έτσι. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό και που έχουμε ακόμα κάποια ελλείμματα είναι πώς θα μεταφέρουμε τις καινοτομίες σε βιομηχανικό επίπεδο, πώς θα κάνουμε τις καινοτομίες προϊόντα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε τώρα για ό,τι θα πρέπει να γίνει για αυτά τα θέματα που αναφέρατε. Ευχαριστώ. Mr. Dartmouth, uh, on behalf of EFD Group. Από την ομάδα Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο κύριος Dartmouth. Θα μιλήσω δεύτερη φορά, ε, εξ ονόματος ενός συναδέλφου που είναι απόν. Κύριε Επίτροπε, αν μου επιτρέπετε, είστε και εντυπωσιακό και η παρουσίασή σας ήταν εντυπωσιακή. Ε, είναι η 37η ερώτηση που σας κάνω και πρέπει τι να σας πω πια. Στο 4-3 πάντως λέτε ότι το εμπόριο θα πρέπει να εξυπηρετήσει ευρύτερους πολιτικούς στόχους. Όπως είπε και ο David Μάρτιν, εδώ έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε προσωπικά. Σας κάνουμε ε, και ερωτήσεις που μπορείτε να τις απαντήσετε προσωπικά. Η ερώτησή μου είναι, εσείς προσωπικά, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ευρωπαϊκές αξίες στις οποίες αναφέρεστε στην ίδια παράγραφο 4.3 και εσείς προσωπικά τι πιστεύετε ότι σημαίνει οι ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί αυτό που έμαθα εγώ στο κοινοβούλιο εδώ είναι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, τα ε, τα εννοεί ο καθένας μας με διαφορετικό τρόπο. Οι προσωπικές μου πεπιθήσεις είναι ότι το μοντέλο της κοινωνίας που έχουμε στην Ευρώπη θα πρέπει να διατηρηθεί. γιατί είναι πολύτιμο. Είναι συνδυασμός ελεύθερης οικονομίας με ευρύτατη κοινωνική προστασία, με εκτεταμένο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και με δικλείδες ασφαλείας σε επίπεδο νομικό. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα για το περιβάλλον θα πρέπει να παίξουμε ηγετικό ρόλο. Στην Κοπεχάγη δεν μπόρεσαν να μας ακολουθήσουν άλλοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω ότι έχουμε και μία αποστολή ε, για την ανάπτυξη και είμαστε ε, ηγέτες σε ό,τι αφορά τη χορήγηση επίσημης ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε σε όλες τις πολιτικές μας. Νομίζω ότι η κοινωνία, η κοινωνία μας βασίζεται σε αξίες και πραγματικά είμαι περήφανος που ανήκω σε αυτή την κοινωνία. Χωρίς μικρόφωνο. Ε, το σημείο μας σας υπονοεί ότι πιστεύετε πως οι εμπορικές πολιτικές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ε, εργαλείο για να εξαχθούν οι ευρωπαϊκές αξίες σε άλλες κοινωνίες. Εγώ έτσι το κατανοώ. Μπορείτε να το διευκρινίσετε. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Η πολιτικοποίηση της εμπορικής πολιτικής ήταν το σήμα κατατεθέν του προκατόχου σας. Και θα ήθελα να εκφράσω την ε, ευχή εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που μας εκπροσωπεί ο Επίτροπος Εμπορίου, κάτι που δεν μας αρέσει, ήθελα να σας πω αυτή η πολιτικοποίηση τη εμπορική πολιτική θα συνεχίσει, θα χρησιμοποιήσει την εμπορική πολιτική για να εξάγεται, εν πάση περιπτώσει, τις αξίες μας. Μπορείτε να το διευκρινίσετε αυτό. Μπορεί και να συμφωνώ με τις αξίες. Αυτό δεν έχει να κάνει. Απλώς, η ερώτηση μου είναι άλλη. Απάντηση. Πρόκειται για αξίες που στηρίζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία και που και που μας εμπνέουν όταν διενεργούμε τις εμπορικές ε, διαπραγματεύσεις. Το εμπόριο είναι και αξία, είναι και αναγκαιότητα. Χρειαζόμαστε το εμπόριο. Είναι θετικό όταν δίνουμε ευκαιρίες στους εταίρους. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αντίφαση. Ε, θα ήθελα να μην αναφερθώ στους προκατόχους μου, αν μου επιτρέπετε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο προκάτοχός μου έκανε μια θαυμάσια δουλειά. Για τον Μάντελσον μίλαγα, έτσι, όχι για την Άστον. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε στο τέλος του χρόνου των ερωτήσεων και θα δώσω το λόγο στον κύριο Φάιρα από την ομάδα των φιλελευθέρων. Θα ήθελα να κάνω ένα ανεπίσημο διάλειμμα να πω χρόνια πολλά στον συνάδελφο για τα γενέθλιά του που έρχεται και περνάει τα γενέθλιά του εδώ στην Ακρόαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε υποψήφι επίτροπε λέει κύριο Στόιρερ. Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ε, ΑΣΕΑΝ Κίνα. Τίθεται το ερώτημα μήπως πρέπει να αλλάξουμε τακτική απέναντι στη Σιγκαπούρη απέναντι στους ε, έξι της ΑΣΕΑΝ, ε, της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ε, πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ασφάλεια πρώτων υλών. Οι πρώτες ύλε είναι σημαντικές για την τεχνολογία, την καινοτομία, ε, για την επιστήμη. Όταν μιλάμε για πρώτες ύλε, έχουμε στο μυαλό μας πρώτα το πετρέλαιο και μετά το φυσικό αέριο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι πολύτιμοι πόροι, όπως είναι το λίθιο για την ηλεκτρική ενέργεια. Και ρωτώ, για σας ως μέλλον επίτροπος για το εμπόριο έχει σημασία αυτό το θέμα και ποια το θεωρείτε σημαντικό για δράση να υπάρξει μια στρατηγική για την εξασφάλιση του ανεφοδιασμού της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας στην Ευρώπη σε τέτοιου είδους πρώτες ύλες. Ε, καταρχάς, χρόνια σας πολλά για τα γενέθλιά σας και από πλευράς μου. Σιγκαπούρη. Καταλήξαμε ότι την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε συμφωνία ελευθερών συναλλαγών με το σύνολο της ΑΣΕΑΝ. Γι' αυτό ακολουθούμε την ε, διμερή προσέγγιση ε, αλλά πολιτικά παραμένουμε προσιλωμένοι στην προσέγγιση την περιφερειακή. Αλλά οι καταστάσει διαφέρουν από χώρο σε χώρα, Προφανώ. Το θέμα των πρώτων υλών είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για 4,5 δις κάθε χρόνο. Με την Κίνα βλέπουμε ότι έχουν ποσοστώσεις, έχουν δασμούς, ελάχιστες τιμές εξαγωγών και χρησιμοποιούν ε, απολύτως και εκμεταλλεύονται την εφευρετικότητά μας. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και σε υψηλότατο επίπεδο οικονομικού διαλόγου με την Κίνα. Αυτό είναι πράγματι κρίσιμο για μας και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και πώς να το πω... Για την ασφάλεια την ίδια τον εφοδιασμό μας. Να έχουμε τα υλικά στις σωστές τιμές και να μην αντιμετωπίζουμε στρεβλές πρακτικές. Με ε, συμπληρωματική ερώτηση. Από την απάντησή σας εκλαμβάνω ότι θεωρείται σημαντικό το θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ποιος θα είναι αρμόδιος επί της ουσίας και είστε πρόθυμος να το συζητάτε και με εμά στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Πρέπει να πω ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ το σύνολο των απαντήσεών σας μέχρι στιγμή. Um, uh, Κοιτάξτε, δεν ξέρω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα είναι η αρμοδιότητα, μα είναι θέματα εμπορικά που πρέπει να συζητούμε εμείς. Και βεβαίως υπάρχει και μια πολιτική πτυχή. Ε, φαντάζομαι ότι όταν... Ε, ε, φτάσουμε σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωση Κίνα, θα συζητηθούν και τέτοια θέματα. Γιατί είναι δύσκολο να αποσιωπήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να θεωρήσει ότι δεν είναι σκεμμένη η πολιτική αυτή. Είναι σκεμμένη και έχει πολιτικούς στόχους. Ε, όχι πάντα εμφανεί, ε, οικονομικούς κυρίως. Παράδειγμα, όταν θα πρέπει εμείς να αγοράσουμε ακριβότερα τις πρώτες ύλες όσο πολλούνται στη χώρα παραγωγής. Αυτό είναι στρέβλωση του εμπορίου. Δεν είναι μια συνειδητή πολιτική στρατηγική, είναι στρέβλωση του εμπορίου οικονομική. Φτάνουν οι ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Ε, είναι πολύ απαιτητικό αυτό ως άσκηση για τον υποψήφιο Επιτροπό μας. και έχει και δικαίωμα σε μια τελική δήλωση προς την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής, εγώ δεν θα κάνω ερώτηση, αλλά θα ήθελα να αναφερθείτε σε ένα θέμα που αξίζει να ακουστεί στην ακρόαση τούτη, που είναι το εξής. Σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει στον καθορισμό της διαπραγματευτικής εντολής ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις. Βεβαίω, σε εσά να να απαντήσετε όπω θέλετε, να κάνετε την τελική σα δήλωση όπω θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω εσά προσωπικά και όλου του συναδέλφου για την ακρόαση αυτή και την ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση που είχαμε με ανοιχτό πνεύμα εκατέρωθεν. εκατέρωθεν. Να απαντήσω πρώτα στην ερώτησή σας. Το Συμβούλιο αποφασίζει την εντολή. Αυτό το ορίζει η Σύνταξη της εγώ δεν μπορώ να το αλλάξω, έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντως αναγνωρίζω ειλικρινά ότι έχετε να διαδραματίσετε πρωταγωνιστικό ρόλο στον καθορισμό της εντολής αυτής. Και είμαι βέβαιος ε, ότι ε, ε, θα εξασφαλίσω να είναι σωστή η διαβούλευση στην Επιτροπή σας. Θα συζητούμε τους στόχους, τους πολιτικούς, τους οικονομικούς, τις μελέτες αντικτύπου που κάθε φορά θα εκπονούμε. Θα έχετε χρόνο και θα το εξασφαλίσω εγώ, θα βεβαιωθώ να έχετε χρόνο για ψηφίσματα και ψηφοφορίες ρητά για τα θέματα και ε, θα τα λάβω σοβαρά υπόψη και δεόντως πάντα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Θα κάνω ό,τι μπορώ δηλαδή, ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ε, σας καταστήσω ισότιμο εταίρος τον καθορισμό της εντολής, όχι μόνο τον καθορισμό, και στην παρακολούθηση της εντολής αυτής κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αλλά πάντα σεβόμενοι ε, με ομικρογιώτα τη συνθήκη της Σαββόνας. Τελικές παρατήρησεις δεν έχω να προσθέσω και πάρα πολλές. Πρέπει να σας πω ότι τα θέματα αυτά ε, καμία φορά είναι πολύ δύσκολα και τα έχω παρακολουθήσει, τα μελέτησα πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι, πραγματικά κάθισα και διάβασα και όταν είσαι 55 ετών δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό. Ε, και το συζήτησα πολύ με τις υπηρεσίες για να δω ε, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ποια είναι η θέση μας και πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε ε, την ανταπόκριση που περιμένετε. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο έτη, εάν επιβεβαιωθεί η θέση μου, θα φροντίσω να κάνω ό,τι μπορώ για το εμπόριο. Αλλά σας είπα ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι για την ευρωπαϊκή ε, κοινωνία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και την ανάπτυξη. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον υπόλοιπο κόσμο να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και μάλιστα η φόρο ανάπτυξη και είναι πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη να το ζήσουμε αυτό. Εάν θέλουμε να είναι βιώσιμο το κοινωνικό μας πρότυπο, Χρειάζεται ανάπτυξη. Και όχι μόνο πώς θα γίνει, αλλά και πώς θα γίνει βιώσιμη και αηφόρος αυτή η ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Thanks. Uh,